Συνάδελφοι, καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, παρακαλώ. Έχουμε την έκθεση για την κίνηση, το μέλλον, δηλαδή, της κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγητής ε, είναι ο κύριος Ούλυρη. ο κύριος Ούγελη, συγγνώμη. Θα σα δώσω το λόγο αυτή αμέσω και στη συνέχεια ο Σκιώδη τις βεβαίω θα πάρει το λόγο ε, για να έχουμε μια μικρή συζήτηση. Θα στήσουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Λοιπόν, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα μιλήσω ουγγρικά, οπότε παρακαλώ τα ακουστικά σας. Ε, Έχουμε εδώ μια εξαιρετικά συναρπαστική έκθεση. Εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών ε, βεβαίως ε, δεν ακολούθησε την κλασική μέθοδο για την έκθεση διότι πρόκειται για ένα πολύ σφαιρικό και πολύ ε, ε, θέμα. Έπρεπε πρώτα να περιορίσουμε λοιπόν το πεδίο, διότι έχουμε μια ανακοίνωση ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκής αφενός, αλλά είναι πολύ ευρύ αυτή η ανακοίνωση. Καλύπτει πολλά πεδία. Εγώ λοιπόν άλλαξα κάπως τη σειρά. Στο Στρασβούργο συναντήθηκα με τους κοιόδης και προσπάθησα να τους εμπλέξω στο ε, στην, στην προσπάθεια που γίνεται ευθύς εξ αρχής, να καθορίσουμε δηλαδή από κοινού ε, τελικά τι θα καλύψει αυτή ε, η εργασία και νομίζω ότι αυτό ήταν καλό θα μας το πούν και οι συγκητές βέβαια διότι μπορέσαμε έτσι να οριοθετήσουμε το έργο μας και ακολουθήσαμε αυτή την προσέγγιση θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους και συγκητές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια πολύ γενική ανακοίνωση, αφορά την κινητικότητα γενικότερα. Ε, προσπαθούμε να καλύψουμε διάφορους τρόπους μεταφοράς ε, και βεβαίως πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονα και ένας σαφής ε, κινητήριος άξονας. Γι' αυτό εμείς δίνουμε εδώ έμφαση στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Γιατί ε, ούτως ή άλλως αυτά τα ζητήματα καλύπτονται και σε άλλες ε, νομοδοτήσει, σε άλλες εκθέσεις. Εδώ, στο κείμενο αυτό, σε πολλέ παραγράφους ε, γίνεται αναφορά, όμως ε, η αυτοματοποίηση, η ψηφιοποίηση, η επίπτωση της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης είναι ακόμα πιο σημαντικά ζητήματα. Γι' αυτό λοιπόν Έχω κάπως ε, συμπτύξει και τον τίτλο της ανακοίνωσης της Κομισιόν στη δική μου έκθεση εδώ. Όπως είπα, είχα μια πρώτη συνάντηση με τους κοιόδους συγητές, ε, συζητήσαμε τις διάφορες προτάσεις ε, που, λάβ, που, που άκουσα από τους συναδέλφους προσπάθησα να τις περιλάβω στο κείμενο βεβαίως δεν υπάρχει χώρος για τα πάντα χωρίζεται σε τρία σκέλη η έκθεση πρώτα μιλάμε για τον αντίκτυπο των αλλαγών στον τομέα της κινητικότητας. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στη μεθοδολογία πώς η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να υποστηρίξουν το όλο εγχείρημα και ε, τρίτον ε, εξετάσαμε πώς ε, από πλευράς κοινωνίας, από πλευράς χρηστών έχουν αλλάξει τα πράγματα στο συγκεκριμένο τομέα. Δεν πρόκειται τώρα να αναφερθώ λεπτομερώς στην ανακοίνωση της Κομισιόν, ούτε στην έκθεση. Να σας πω μόνο λίγα λόγια. Η πρόταση, η πρόταση της αναφέρεται εξαντλητικά σε όλες τις προτάσεις ε, των προηγούμενων ετών για το πώς ε, η κινητικότητα θα εξελιχθεί στο μέλλον. Η ιδέα της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η κινητικότητα θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική, ε, να υπάρχει συνδεσιμότητα και να βρίσκεται η Ευρώπη στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Αυτά είχα να πω, διότι νομίζω πως είναι σημαντικό να ακούσουμε και τους εκπροσώπους των λοιπόν πολιτικών ομάδων. Σε γενικές γραμμές πάντως το που μπορώ να πω είναι ότι εμείς συντάξαμε ένα κείμενο το οποίο ακολουθεί μια σφαιρική προσέγγιση δεν χανόμαστε στις λεπτομέρειες, θέτουμε συγκεκριμένους στόχους, μιλάμε για μια προσβάσιμη ασφαλή, ένα προσβάσιμο ασφαλή τομέα μεταφορών, μιλάμε για την ανάπτυξη και κυρίως για την προσβασιμότητα για τους χρήστες. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ουρή. Κύριε Δεγκράντε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή αλλά και τους κοιόδης εισηγητές. Θα είμαι σύντομος, όπως ήταν και ο εισηγητής. Θέλω να ευχαριστήσω πάντως τον εισηγητή. Όντως έγινε μια συνάντηση άτυπη και προσπαθήσαμε από κοινού να οριοθετήσουμε αυτή την έκθεση διότι ήταν πολύ γενικόλογη η προσέγγιση της Κομισιόν είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε ε, διότι καλύπτει πολλά και διάφορα η έκθεση αυτή και έπρεπε να το υιοθετήσουμε και το κάναμε νομίζω αυτό με έξυπνο τρόπο. Το έκανε έξυπνα ο εισηγητή και θέλω να τον ευχαριστήσω. Διότι σε αυτή την έκθεση πρωτοβουλία ε, έχουμε οδηγηθεί τώρα σε ένα ισορροπημένο και λογικό κείμενο. Είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε όπω είπα και ε, νομίζω ότι αποτυπώνονται οι απόψει μα στο κείμενο και γι' αυτό ευχαριστώ τον εισηγητή. Πιστεύω ότι οι απόψει των κοινών εισηγητών ε, ελήφθησαν υπόψη ότι έκανε μια σύνθεση, μια πραγματική σύνθεση ο εισηγητή. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, μα αφορά όλου. Είναι σχεδόν μελλοντολογία βέβαια αυτό που κάνουμε, αλλά δεν κάνει κακό αυτό. Να κοιτάζουμε και λίγο προ το μέλλον, διότι εξετάζουμε και το πακέτο, ε, εξετάζουμε μάλλον τα, τα καθημερινά, αλλά Έχουμε τι νέε τεχνολογίες, ε, τις έξυπνες τεχνολογίες, την ψηφιοποίηση, όλα αυτά είναι ένα φαινόμενο, αποτελούν ένα φαινόμενο το οποίο είναι χωρίς επιστροφή. Και αυτό θα επηρεάσει την κινητικότητα, του νέου τρόπου μεταφοράς στο μέλλον. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μια συμβίωση, να υπάρχει ένας ε, πολυτροπικό πολυτροπική προσέγγιση ότι φορές μεταφορές. Ως και ως συγητές βέβαια, ως και ως ε, θα υποβάλω μια σειρά από τροπολογίες ε, που αφορούν την ασφάλεια, που αφορούν την νομιμότητα αυτών των νέων τρόπων μεταφοράς, ε, την νομική ευθύνη, αλλά και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τα συζητήσαμε αυτά ε, σε γενικές γραμμές και θα κάνουμε και κάποιε, θα βάλουμε κάποιε τροπολογίε για τα ζητήματα που μα ανησυχούν περισσότερο. Φαντάζομαι ότι όλοι θα συμμεριστούν αυτέ τι ανησυχίε και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε ελεύθερα ε, για να ε, αυτέ αυτές τις πτυχές ε, που αφορούν το μέλλον. Το μέλλον όμω είναι ήδη σήμερα, είναι πολύ κοντά και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Εγώ έχω κάθε πρόθεση να συνεργαστώ στα πλαίσια αυτής της ε, έκθεσης πρέπει τα νέα και τα παλαιά, οι νέοι και παλαιοί τρόποι μεταφοράς να μπορέσουν να συγκεραστούν, να συνυπάρξουν. Η συνεταιριστική οικονομία επίσης, ε, ε, στην οποία βέβαια βάζουμε μέσα πολλά πράγματα ε, και δεν μπορεί να είναι μια ζούγκλα, δεν μπορεί να, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει εκεί, πρέπει να υπάρχει μια ρύθμιση, να υπάρχουν σαφείς κανόνες του παιχνιδιού, να μην παρεμποδίζουμε την καινοτομία αλλά να σεβόμαστε ταυτόχρονα και τα κεκτημένα δικαιώματα. Αυτά είναι οι δύο βασικοί άξονες, ε, διότι έχει σημασία αυτό για λόγους ισοτιμίας, να μην παρεμποδίζουμε το μέλλον που έρχεται, αλλά να σεβόμαστε αυτά που υπάρχουν. Θα πρέπει λοιπόν η νέα νομοθεσία να μην οδηγεί απλώς ε, στο να αποφασίζονται τα ζητήματα αυτά στα δικαστήρια, διότι αυτό συμβαίνει συχνά. Ε, δεν παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις, ε, ρυθμίσεις δεν υπάρχουν και τελικά έχουμε διαδοχικές ε, αποφάσεις δικαστηρίων οι οποίες μάλιστα συχνά είναι αντικρουόμενες μεταξύ τους και δεν είναι αυτό το, ένα, μια κατάσταση την οποία μπορούμε να αφήσουμε να συνεχίζεται ως πολιτική ηθήνοντες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ντεγκράντε. Ο κύριος Βαν Μίλτεμπουργκ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω κι εγώ στη μητρική μου. Καταρχάς να ευχαριστήσω κι εγώ τον εισηγητή για το σχέδιο κειμένου για το μέλλον της ε, κινητικότητας και των μεταφορών στην Ευρώπη. Είναι παρόμοια τα σχολεία μου με αυτά που ε, ανέφερε και ο εισηγητή ότι έγιναν στην συνάντηση με τους σκιώδει εισηγητέ. Βεβαίω δεν είναι εύκολο να ε, υπάρξει μια τέτοια στρατηγική έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποια συγκεκριμένα επιμέρους ζητήματα και αυτό το έκανε πολύ καλά ο εισηγητής. Ψηφιοποίηση, καινοτομία, βιωσιμότητα, ασφάλεια. Όλα αυτά είναι πολύ ουσιώδη σημεία. Τώρα για τη βιωσιμότητα. Έχουμε πολλές ευκαιρίες για τον τομέα των μεταφορών, για το μέλλον και για την οικονομική ανάπτυξη μέσω ε, χρήσης καθαρών τεχνολογιών, αλλά και δουλεύοντας επί τη βάση του ορυπαίνων πληρώνει αυτή τη αρχή. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ε, ισοτιμία όπλων ουσιαστικά μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφορών. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα, η Ευρωβινιέτα και άλλα, τα οποία θα μπορούσαμε ίσως να μελετήσουμε, γιατί ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό από άποψη βιωσιμότητας. Ένα δεύτερο σημαντικό είναι η ψηφιοποίηση και η καινοτομία. Η ε, γνωμοδότηση μπαίνει σε λεπτομέρειες ως προς αυτό το θέμα, ε, καινοτόμος τεχνολογία για πράσινες μεταφορές. Ε, συνδεδεμένα αυτόματα οχήματα. Ε, επίσης ένα θέμα σημαντικό και πρέπει να υπάρξει και πρόοδο ό,τι αφορά την τυποποίηση σε τεχνικό επίπεδο και πρέπει να έχουμε υπόψη βεβαίως και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η προστασία λοιπόν των δεδομένων και η ιδιωτικότητα αναφέρεται από τον εισηγητή και χαίρομαι πολύ που το έκανε, που το ανέφερε στην εκθεσή του, γιατί όντω είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό. Επίση, η καινοτομία δεν έχει να κάνει μόνο με την πρόοδο τη τεχνολογία, έχει να κάνει και με την κοινωνική ε, πρόοδο. Πώ μπορούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ίσω νέε δεξιότητε στην ε, αγορά εργασία, έτσι ώστε οι πολίτε να μπορούν να βρουν πιο εύκολα δουλειά στον τομέα αυτό. Το λέει και, σε αυτό, και στην έκθεση του αυτό Και επίση η ασφάλεια, Πρόεδρε. Πρέπει να βελτιωθεί γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα στην Ευρώπη και η Ευρώπη πραγματικά πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα της ασφάλειας. Αν θέλουμε, αν κάποια στιγμή αποκτήσουμε αυτόματα οχήματα, που θα μοιράζονται τους δρόμους με οχήματα που δεν είναι ε, αυτόματα, αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη, ας πούμε, σε τούνελ ή σε άλλα σημεία των ε, ε, δρόμων. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτού. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τρόποι με, με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η έκθεση, αλλά γενικώ είναι πολύ καλή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δελοντέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ όπως και οι προλαλήσαντες θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετική αυτή η έκθεση διότι πραγματικά μας μιλάει για το μέλλον. Για αυτά που θα γίνουν το μέλλον. Το εκτιμάμε ιδιαίτερα και θεωρούμε ότι πρέπει να καθορίσουμε προτεραιότητες να ενθαρρύνουμε τους καταναλωτές ε, να στραφούν προς οχήματα πιο οικονομικά, πιο πράσινα. Η αρχή του ρηπαίνοντος που πληρώνει είναι εξαιρετική. Επίσης υπάρχει το σύστημα bonus μάλους το οποίο είναι σημαντικό. Αυτό μπορεί να ε, παροτρύνει τους καταναλωτές να αγοράσουν πιο καθαρά οχήματα. Θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό να λαμβάνει κανείς ε, κάποιον έπαινο, κάποιον πόνου όταν ε, αγοράζει ένα καθαρό αυτοκίνητο. Ποιος θα το πληρώσει όμως ε, όλη η κοινωνία. Όχι, θα το πληρώσουν αυτοί που έχουν μάλους, δηλαδή αυτοί που αγοράζουν ε, οχήματα τα οποία ρηπαίνουν. Έτσι θα υπάρχει μια ισορροπία. Όσοι αγοράζουν καθαρά οχήματα θα ενθαρρύνονται λόγω των οικονομικών κινήτρων, τα οποία θα καταβάλλονται από αυτούς που αγοράζουν βρώμικα οχήματα, οχήματα που ρηπαίνουν. Επίσης ε, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι οι τιμέ πρέπει να είναι λογικέ όταν αναφερόμαστε στη χρήση των ε, δρόμων διότι όταν ε, υπάρχει κυκλοφορία και συμφόρηση δημιουργείται τεράστια ρήπανση και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πολλά προβλήματα θα λυθούν με τα αυτόνομα οχήματα γιατί ενδεχομένως στο μέλλον θα έχουμε λιγότερες θέσεις στάθμευσης οπότε οι πόλεις μας θα έχουν λιγότερη κίνηση. Θα είναι πιο ευχάριστε στη διαβίωση. Ε, τα καφέ θα μπορούν να βγάζουν τραπέζια στα, τραπέζια, στα πεζοδρόμια χωρί να υπάρχει μόλυνση. Ευχαριστούμε κύριε Ντελόντα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι... Συγγνώμη, δεν είδα. Παρακαλώ, Βήμ. Κυρία Πρόεδρε, Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω δύο σχόλια για τα όσα είπε ο συνάδελφος ο κ. Λουίδε Γκράντες. Υποστηρίζω τα όσα είπε και τα όσα είπε και ο κ. Βαν για την ποιότητα τη ε, πρόταση, αλλά για να μην ειλικρινή, εδώ λείπει κάτι. Λείπει μια ε, ιδεολογία που είχαμε παλιότερα που αφορά τη διατροπικότητα και την αλλαγή τρόπου μεταφορών. Αυτό μου θυμίζει το κείμενο σε της, ε, της περασμένης εβδομάδας, το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό κείμενο. Μεν, παρόλα αυτά, εξακολουθούν να κυκλοφορούν χιλιάδες ε, φορτηγά και για να έχουμε μια έκθεση που να καλύπτει τα πάντα, όπως αναφέρεται στη Λευκή Βιβλό του 2011, θα ήθελα να έχουμε τις λέξεις «model shift και intermodality μέσα στην έκθεση ως βασική έννοια του κειμένου μαζί με την ιδέα της ε, κινητικότητας ως υπηρεσία. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον εισηγητή, συμφωνείτε μαζί μου, ενδεχομένως όχι, αν όχι θα μπορούσαμε να υποβάλουμε κάποια τροπολογία ενδεχομένως. Ευχαριστούμε ο κύριος Τελίνσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τίποτα από όσα υπόθηκαν για την ποιότητα της έκθεσης και για τα βασικά της στοιχεία, αλλά κάποιος αναφέρθηκε σε μια ε, στρατηγική ε, προοπτική. Αν έχουμε μια αρχική έκθεση με στρατηγική προοπτική, θα πρέπει να γίνει και μια αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης, του σημερινού οικοσυστήματος. Άνευ των οποίων ε, δεν θα είναι πλήρης η έκθεση. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μερικές προτάσεις. Δεν θέλουμε απλά να πούμε κάποιες γενικολογίες, να αξιολογήσουμε πλήρως το σημερινό σύστημα για να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ε, στους ε, συνομοθέτες. Αυτή είναι η σύντομη παρατήρηση, αλλά θα ήθελα να τη λάβει υπόψη ο σε Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τέλισκα. Κύριε Ερτούγκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ είμαι της άποψης ότι η έκθεση αυτή θα μπορούσε να συμβάλλει στο να μπορέσουμε να προλάβουμε ίσως τις μελλοντικέ τάσεις ε, όσοι ε, γνωρίζουν την κατάσταση στην ε, Γερμανία ξέρουν ότι σήμερα θα αποφασίσει το ανώτερο δικαστήριο αν στο εγγύς μέλλον στην Γερμανία θα πρέπει να υπάρξουν απαγορεύσεις για φορτηγά τα οποία δεν τηρούν τα όρια των εκπομπών αερίων για να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι η κινητο... βεβαίως η κινητοποίηση είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί ε, όλοι το έχουμε υπόψη μας αυτό, αλλά στην έκθεση αυτή θεωρώ ότι νομίζω ότι έχουν επιλεγεί τα σωστά κίνητρα. Υπάρχουν οι παρατηρήσεις ε, για την ε, Λευκή Βίβλο από, την, το 2011 που μπορούμε να την ενισχύσουμε βεβαίως, είναι σωστά ωστόσο, αλλά να μην ξεχνούμε το εξή. Από το 2011, 7 χρόνια έχουν περάσει σχεδόν και έχουν γίνει πολλά σε αυτά τα 7 χρόνια. Έχουμε ζήσει το σκάνδαλο με, τα, ε, με τις εκπομπές αερίων που νομίζω ότι ε, επηρέασε πάρα πολύ την, ε, την αλυσίδα παραγωγής σε όλο τον κόσμο. Κυρίως βεβαίως στις βιομηχανικές χώρες. Μετά έχουμε την νομοθεσία για τα φορτηγά και τις εκπομπές αερίων. Έχουμε το δεύτερο πακέτο ε, για, τα, για την κινητικότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία τώρα θα τα μεταφέρουμε σε νομοθεσία. Αυτό λοιπόν μας δείχνει ότι το θέμα των μεταφορών πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Και επίσης πιστεύω ότι όταν μιλούμε για την ψηφιοποίηση, δεν θα πρέπει να λέμε ότι μιλούμε μόνο για την προστασία των δεδομένων. Βεβαίω και αυτό χωρί καμία αμφιβολία. Ω ε, σοσιαλδημοκράτη βεβαίω θα, το, θα το υπογραμμίσω αυτό, αλλά μιλούμε και για άλλα πράγματα. Η ψηφιοποίηση θα τα αλλάξει όλα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ε, θα είναι πολύ δύσκολο αυτό η ε, πολιτική εκπαίδευση σχετικά θα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και μάλιστα σε κάποια κράτη των κρατηδίων. Οπότε θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα άτομα αυτά που δεν θα βγουν στη σύνταξη τα επόμενα 15 χρόνια θα πρέπει να κινητοποιηθούν ώστε να κατανοήσουν τι θα σημάνει αυτή η ψηφιοποίηση, πώς θα τη χρησιμοποιήσουν, πώς θα χρησιμοποιήσουν τη νέα τεχνολογία την οποία ούτε μπορούμε να φανταστούμε καν σήμερα και πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν τις ε, αλυσίδες ε, παραγωγής. Αν υπάρχει μεγάλη ε, ας πούμε, παραγωγή από την Γερμανία που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη παραγωγή γιατί έχει καλά αποτελέσματα θα πρέπει να, να δούμε τι θα γίνει και με τα κέρδη των βιομηχανιών. Γιατί και, αυτοί, και αυτές θα πρέπει να κάνουν το μεγάλο βήμα προς την ηλεκτροκίνηση. Βεβαίω υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι σε πέντε χρόνια όλα θα έχουν περάσει σε ηλεκτροκίνηση. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Θα έχουμε μια μεταβατική φάση πρώτα που αν πάει καλά μπορεί να κρατήσει και 10-15 χρόνια. Αν δεν πάει καλά μπορεί να κρατήσει πάνω από 20 χρόνια. Αλλά αυτή η μεταβατική περίοδος θα μπορούσε με αυτά τα υβριδικά μοντέλα, με το power to gas κτλ. να ξεπεράσει τα προβλήματα. Και ως τελευταία φράση να πω ότι αν όντω θέλουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο αυτό της ηλεκτροκίνησης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η βιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία συγκεκριμένα, θα μπορεί να πουλήσει και τα αυτοκίνητά τη. Ίσως να ακούγεται και λίγο τρομακτικό αυτό, αλλά μόνο η, η αυτοκινητοβιομηχανία δεν μπορεί να έχει μόνο αυτό το καθήκον και δεν είναι μόνο δικό της, καθήκον. Πρέπει να δημιουργήσουμε και οικοσυστήματα τα οποία θα μπορούν να καλύψουν τα, την ηλεκτροκίνηση. Αυτό προς τη στιγμή δεν υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να κατασκευάσουμε ευφυείς e δρόμους, ευφυεί e δίκτυα Έχουμε και τα ε, θέματα της ε, παραγωγής και των αδειών και βεβαίως οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ πιο αυστηρές ως προς αυτό το τομέα. Οπότε όλο αυτό το περίπλοκο θέμα δεν μπορούμε μόνο να το βλέπουμε από τη θεώρηση της έξυπνης νομοθεσίας που γράφουμε. Η αλλαγή πρέπει να γίνει πραγματικά σε όλα τα επίπεδα. Ε, πριν από 10 μέρες έκανα εγώ μια σχετική πρόταση με το European Clean Mobility Fund. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες ώστε οι ε, υποδομές να είναι διαθέσιμες έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Και στο σημείο αυτό ε, έκλεισε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνω να, ότι είναι λάθος να υποβάλει μόνο μία ανακοίνωση. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένη νομοθεσία δεσμευτική που να βασίζεται σε δεδομένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μάσνερ, έχετε το λόγο. Μια σύντομη παρατήρηση. Η έκθεση είναι καλή και είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με την κινητικότητα στο μέλλον. Για την ψηφιοποίηση θέλω και εγώ να πω κάτι που όντω θα αλλάξει πολλά όταν θα υπάρξει και όταν θα είναι πολυτροπική. Εμείς στο, ήμασταν στο πρωινό της ε, Reform from Europe και ήταν και εκπρόσωποι της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρόντες, ένας από τον οποίο είναι εδώ μάλιστα τώρα, και μπορώ να σας πω τι σχεδιάζει η Κομισιόν, γιατί η ψηφιοποίηση είναι γνωστή. Ε, μιλάμε για, την, ε, για ολόκληρη την αλυσίδα των ε, οχημάτων. Όχι όμως μόνο για τα οχήματα, μιλούμε για τα φορτηγά, μιλούμε για τα τρένα, μιλούμε για τα πλοία. Η ψηφιοποίηση θα αφορά όλους τους κλάδους. Οπότε εξαρτάται και από, την, από το τι θα έρθει από την Κομισιόν, εξαρτάται και από του πολίτε που θα τη χρησιμοποιήσουν και πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικότητα ε, αυτάρκεια ό,τι αφορά την ενέργεια και τη χρήση ενέργεια και όλα τα σημεία αυτά θα μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε. Γι' αυτό Εμεί, από τη δική μα την πλευρά, από το Βούλιο από κοινού με την Κομισιόν θα πρέπει αυτά να τα προωθήσουμε. Αλλά παρόλα αυτά η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μάιστα, Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Ωραία, να μιλήσω κι εγώ λοιπόν. πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική έκθεση, διότι πρέπει να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα για το μέλλον της κινητικότητας στην Ευρώπη. Αυτές οι λέξεις σημαίνουν κάτι. Η λέξη πρόγραμμα, η λέξη μέλλον. Τι θα συμβαίνει στο μέλλον. Θα είναι τελείως διαφορετικό, διαφορετικά τα πράγματα σε επίπεδο κλίματος. Έχουμε διακυβεύματα σημαντικά. Η COP21 μας λέει ότι ο τομέα των μεταφορών δεν μειώνει ε, τις, εκπομπές. Πώς θα επιλύσουμε στο μέλλον αυτήν την ασθένεια του 21ου αιώνα, ε, τη μόλυνση. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα Ηνωμένα Έθνη. Η μεγάλη ασθένεια του 21ου αιώνα είναι η μόλυνση. Αυτό σημαίνει 500.000 πρόωροι θάνατοι ε, στη χώρα μου, παραδείγματο, χάρη τη Γαλλία. Κάτι άλλο που έχει σημασία, δεν το έχουμε πει επαρκώ. η κινητικότητα στο μέλλον πρέπει να είναι προσβάσιμη για όλους και για τα άτομα με αναπηρία αλλά και για τα άτομα που δεν έχουν τα μέσα αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν επισφάλεια σε παιδοκινητικότητα. άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση δηλαδή στα μέσα μεταφορών επειδή ε, δεν υπάρχει κάτι κοντά στο σπίτι τους ή επειδή δεν έχουν τα χρήματα για να πληρώσουν στο μέλλον λοιπόν πρέπει ε, η κινητικότητα να μπορεί να καλύπτει όλους τους πολίτες το τρίτο σημαντικό στοιχείο. Μια κινητικότητα η οποία να διέπεται από συνδεσιμότητα. Βεβαίω μιλάμε εδώ και καιρό για το αυτόνομο αυτοκίνητο, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα ω εκεί. Αυτόνομο αυτοκίνητο σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε προς, προς πειραματικές προσπάθειες. Ο κ. Βαν Μίλτεμπεργκ προηγουμένως ανέφερε κάτι πολύ σημαντικό. Μίλησε για τα δεδομένα. Ε, Πολύ σημαντικό ζήτημα και όχι μόνο, διότι έχουμε και το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Έχουμε το θέμα της ευθύνης στα πλαίσια του αυτόνομου αυτοκινήτου πάντα. Επίσης ε, πρέπει εδώ να καλύψουμε κάποια χάσματα και το πρόβλημα με τα χάσματα είναι ότι δεν έχουμε όλοι ε, στην Ευρώπη ψηφιακό ε, ε, έξυπνο τηλέφωνο ούτε ψηφιακή σύνδεση και επίση πώ θα συνδέσουμε τα διάφορα εδάφη, διότι η κινητικότητα σημαίνει διάδραση, αν θέλουμε να υπάρχει ε, συνοχή μεταξύ των εδαφών. Επίση, αναφερθήκατε στο θέμα της ασφάλειας, ε, αυτό το μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να είναι, θα πρέπει να είναι στην καρδιά τη συζήτηση και έχουμε και αυτή τη νέα οικονομία, την συνεταιριστική, ε, η οποία είναι διαφορετική από την οικονομία με τις πλατφόρμες και πρέπει αυτή να την πλαισιώσουμε Ιδάλω ε, ο ένα θα μπαίνει στην οικονομία με τι πλατφόρμε, ο άλλο στην συντεστική οικονομία. Θα πρέπει να περιμένουμε να πάρουν, να πάρουν αποφάσει σε επίπεδο δικαιοσύνη για να αποσαφινιστούν τα πράγματα. Και τέλο, αυτό το είπε και ο κύριο και το είπε ο κύριο Έρτουγκ, η κινητικότητα στο μέλλον θα πρέπει να περιλαμβάνει μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική για την μετάβαση της αυτοκινητομηχανίας, για την ε, μετάλλαξή της. Δεν γίνεται πια να προχωρήσουμε με ρηκτά καύσιμα. Είναι εκατομμύρια εργαζόμενοι που θα πρέπει να, βρουν, να μια άλλη δουλειά. Είναι πολύ, ε, πολύ μεγάλο το έργο που μας περιμένει. Εγώ λοιπόν θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες σε σχέση με αυτή τη φιλοδοξία και σε σχέση και με την αλλαγή του δόγματος, έτσι, διότι η κινητικότητα δεν είναι πλέον κάτι το ατομικό, δεν θα είναι στο μέλλον. Θα βασίζεται ε, στο πώς ε, θα μοιραζόμαστε τα πράγματα, διότι το αυτόνομο αυτοκίνητο δεν θα ανήκει σε έναν άνθρωπο, θα το μοιραζόμαστε. Θα πρέπει από εκεί πέρα να δούμε πώς όλα αυτά θα τα πλησιώσουμε. Κάποιος παίρνει ένα τρένο στη συνέχεια ε, ποδήλατο και μετά με τα πόδια. Πώς το διευκολύνουμε αυτό και πώς ε, αυτό το πλαίσιο προστατεύεται και πλαισιώνεται και, και ρυθμίζεται μάλλον. Ε, η Ιζαμπέλ Βαντόρν έχει το λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Θα μιλήσω γαλλικά, κυρία Πρόεδρε. Εμείς δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο να κάνουμε για το σχέδιο έκθεσης ούτε για τις ε, παρεμβάσεις που ακούσαμε σήμερα. Ε, κάποιες πληροφορίες απλώς να σας δώσω. Ε, εδώ δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια. Θα γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει σε λίγες εβδομάδες την άνοιξη, ελπίζουμε να μπορούμε να παρουσιάσουμε το τρίτο πακέτο κινητικότητας που θα αφορά και ζητήματα οδικής ασφάλειας. Θα γνωρίζετε επίσης ότι ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει και το πακέτο για τα δεδομένα όπου ελπίζουμε να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε για να επιτεθούν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν, που αναφέρθηκαν σήμερα μεταξύ άλλων. Ε, το κοινωνικό σκέλος και το εκπαιδευτικό σκέλος έχει και αυτό τη σημασία του Αναφερθήκατε σε μια μελέτη που βρίσκεται να εξελίξει για να απαντήσω στο αίτημά σας ε, για μια ενδιάμεση έκθεση. Από ό,τι φαίνεται κάποιες πληροφορίες ε, θα μπορέσουμε να τις μοιραστούμε μαζί σας όταν θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Σε κάτι άλλο το οποίο αναφέρετε στην έκθεσή σας είναι το θέμα της υπαίθρου για την κινητικότητα. Χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε σύντομα να υπογράψουμε ε, το, τη σχετική σύμβαση για να γίνουν οι εργασίες σχετικά με την κινητικότητα στην Ήπεθρο. Χαιρόμαστε που η Γενική Διεύθυνση Τραν έδωσε όθηση σε αυτό το εγχείρημα και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω, ε, δεν είπατε βέβαια, δεν είπε κανείς αυτή τη λέξη, αλλά η κυρία Μπούλτς θέλει να ε, προωθήσει το θέμα των πολυτροπικών ε, μέσων μεταφοράς, ε, τρόπων μεταφοράς. Όντως η κινητικότητα δεν θα είναι ατομική, θα χρησιμοποιούμε πολλούς, πολλά μέσα, πολλούς τρόπους μεταφοράς και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Νομίζω ότι κάλυψα τα διάφορα ζητήματα σχετικά με την Γενική Διεύθυνση MOVE τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος, ο εισηγητής, ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μελή της Επιτροπής Τραν, άκουσα τις διάφορες απόψεις με μεγάλη μου χαρά. Όσοι από εσάς καταφέρατε να έρθετε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις Βρυξέλλες, ε, βλέπετε την απόδειξη ότι είναι αναγκαίο να ασχοληθούμε με το μέλλον των μεταφορών είτε μιλάμε για αστικές είτε για αγροτικές περιοχές. Οι αστικές διαδρομές παρουσιάζουν όλο και μεγαλύτερη συμφόρηση και τα πράγματα είναι δεινά για το περιβάλλον όπως τα βλέπουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Έτσι λοιπόν πολλές είναι οι με τις οποίες θα πρέπει να ασχοληθεί αυτή η έκθεση. Ωστόσο δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα πάντα μέσα από μια έκθεση. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας ζητήσω να μην υποβάλλετε τις κλασικές, τις συνήθεις τροπολογίες. Σας παρακαλώ να μου δώσετε, να μου υποβάλλετε έξυπνες ιδέες για αυτή την κοινή μας έκθεση. Ε, θα μπορέσουμε λοιπόν έτσι να εργαστούμε, ε, να επεξεργαστούμε την έκθεση αυτή μέχρι να συλλέξουμε τις πιο σοφές ιδέες των μελών αυτής της Επιτροπής. Έτσι στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε αυτή την έκθεση ως ένα κοινό θησαυρό, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για τους πολίτες γενικότερα. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε μία έκθεση την περασμένη εβδομάδα και με τους κοιόδης εισηγητές αποτελούσε ε, το αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειά. Ε, όπως είπε και ο Βήμα Βαντενκάμπα, ε, σχετίζονται οι δύο αυτές εκθέσεις μεταξύ τους. Αντιλαμβάνομαι και αυτά που είπε η Πρόεδρος Μέσα στις επόμενες εβδομάδες λοιπόν θα ήθελα να συλλέξω και να εντάξω όσο το δυνατόν περισσότερες από τις απόψεις, από τα σχόλια που ακούσαμε στην έκθεση. Σας ευχαριστώ. Θα κάνω τις σκληρότερες δυνατές προσπάθειες για να παρουσιάσουμε μια καλή έκθεση. Ευχαριστούμε κύριε Λερή. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 9η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι. Και συνεχίζουμε με το επόμενο σημείο τον τουρισμό για λόγους υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τομάς Μενίλ. Πού βρίσκεστε κύριε Τομάς Μενίλ? Είστε εδώ, δίπλα μου μάλιστα. Καλημέρα. Allez-y, prenez place. Alors, vous allez nous Καθίστε, θα μας προσφέρετε τη μελέτη για τον τουρισμό για λόγους υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 10 λεπτά. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τα μέλη, τα οποία το επιθυμούν. Και μετά θα σας ζητήσω κύριε Μενίλ να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία στην Επιτροπή σας να παρουσιάσω αυτή τη μελέτη για τον τουρισμό για λόγους υγείας. Εργάζομαι στο κέντρο αηφορίας τουρισμού και μεταφορών των κάτω χωρών στο Πανεπιστήμιο της Μπρέντα. Αρχικά θα σας δώσω κάποιους ορισμούς και μετά κάποια νούμερα. Θα σας παρουσιάσω τις πολιτικές ε, που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό και σε περιφερειακό επίπεδο. Θα κάνουμε μια ανάλυση SWOT ε, θα προτείνουμε δύο σενάρια και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα και συστάσεις. Πρώτα απ' όλα, ε, πώς ορίζεται ο τουρισμός για λόγους υγείας. Ε, τον αναφέρουμε και ως μορφές τουρισμού που εστιάζονται στη, φυσική, στη σωματική υγεία, στην πνευματική και ψυχική ευημερία. Ουσιαστικά είναι μια γενική έννοια ο τουρισμός για την υγεία Ουσιαστικά έχουμε τον ιατρικό τουρισμό, άνθρωπου που πάνε σε μια άλλη χώρα για ιατρικούς λόγους. Ο τουρισμός ευεξία είναι για την ενίσχυση της προσωπικής υγείας και τη ευημερία βάσει κάποιε δραστηριότητες και ο τουρισμός σε ιαματικά κέντρα αφορά τη χαλάρωση, τη θεραπεία, την ομορφιά μέσω της παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν ο τουρισμός για λόγους υγείας είναι η γενική ορολογία, ο γενικός όρος ε, που χωρίζεται σε ιατρικό τουρισμό, τουρισμό για λόγους και τουρισμό σε ιαματικά κέντρα. Αν δούμε κάποια νούμερα θα παρατηρήσουμε ότι ο τουρισμός για λόγους υγείας δεν είναι τόσο μεγάλο ε, μερίδιο των συνολικών τουριστικών ταξιδιών. Είναι μόλις το 4,3%. Είναι περισσότερο εγχώριο φαινόμενο παρά διεθνές. Αν δείτε ποια είναι τα έσοδα από τον τουρισμό για λόγους υγείας ε, του εγχώριου και του διεθνούς ε, θα παρατηρήσουμε ότι ε, χωρίζεται σε διάφορες χώρες. Τα τρία τέταρτα ουσιαστικά αντιστοιχούν σε πέντε χώρες. Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία και Σουηδία. Πάμε να δούμε κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες για τις ευρωπαϊκές πολιτικές βλέπουμε ότι αυτές για την κινητικότητα των ασθενών ε, είναι υπαρκτές ως πολιτικές, αλλά όχι συγκεκριμένα για τον τουρισμό για λόγους υγείας, παρότι υπάρχει κάποια στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υπάρχει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά υπάρχουν πολλά διαφορετικά εθνικά, φορολογικά, οικονομικά και νομικά καθεστώτα μεταξύ των κρατών μελών. Περισσότερη εστίαση σε εθνικέ και περιφερειακέ πολιτικέ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πολιτικέ οι οποίε έχουν αναπτυχθεί στα κράτη-μέλη αφορούν περισσότερο την υποστήριξη της συνεργασίας ε, στο πλαίσιο ε, τμήματων ε, κατηγοριών συγκεκριμένων ή ενδιαφερομένων που προσπαθούν να προωθήσουν αυτόν τον τουρισμό να τον παρουσιάσουν σε διάφορες περιοχές με συγκεκριμένο τρόπο, να τον προωθήσουν και αυτό έχει να κάνει και με την διασυνορική κινητικότητα των ασθενών. Αν δούμε μετά την ανάλυση SWOT, ας δούμε πρώτα απ' όλα τα ισχυρά σημεία. Όπως βλέπουμε παράγει σημαντικό εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο τουρισμός για λόγους υγείας. Υπάρχει μεγάλη ιστορία, υπάρχει κάποια ανεπτυγμένη, υπάρχουν ανεπτυγμένες υποδομές σε πολύ καλό σημείο. Η οδηγία θα μπορούσε να αποτελέσει πολύ καλή αφετηρία και επίσης η ποιότητα θεωρείται ότι είναι αρκετά υψηλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δύναμα σημεία είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί, η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων για τον τουρισμό υγείας, η αγορά επίσης δεν είναι ιδιαίτερα ρυθμιζόμενη και δεν έχει προωθηθεί αρκετά ο τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευκαιρίες που παρουσιάζει ο τομέα, πολλοί είναι οι πολίτε που επιθυμούν να ταξιδέψουν για ιατρική φροντίδα, χρήση ICT και πόρων ε, διαδικτυακών για τη σύνδεση των καταναλωτών και η γύραση του πληθυσμού. Όλα αυτά προσφέρουν ευκαιρίε για έρευνα και ανάπτυξη. Ως απειλέ, ε, παρατηρούμε την έλλειψη τη ευαισθητοποίηση του γνώση της γνώσης του κοινού όσον αφορά την οδηγία. Επίση υπάρχει πολύ αρνητική παρουσία στον τύπο όταν τα πράγματα δεν πάνε όπω ε, είναι επιθυμητό και επίση οι κυβερνήσει φοβούνται ότι οι πολίτε θα εγκαταλείψουν τα εθνικά συστήματα υγεία ε, για τον ιατρικό τουρισμό, προ όφελο του ιατρικού τουρισμού και τη κινητικότητα των ασθενών. Ας δούμε τώρα τα πιθανά σενάρια αυτά είναι περισσότερο θεωρητικά. Το σενάριο ανάπτυξης του τουρισμού για λόγους υγείας, όπου λέμε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές ε, θα οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη του τουρισμού για λόγους υγείας, αλλά και οι ιδιωτικές επενδύσεις ε, όλο ένα αυξάνονται για τα ΣΠΑ και για τους προορισμούς ευεξίας ε, εφόσον αφαιρεθεί και η σχετική νομοθεσία ότι θα υπάρξουν εταιρικές σχέσεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη της αγορά και θα ανοίξουν και τα εθνικά συστήματα υγείας. Είναι ένα θεωρητικό σενάριο αυτό και αποτελεί τη μία ε, εικόνα που μπορούμε να έχουμε. Υπάρχει το άλλο σενάριο της ζωτικότητας του τουρισμού της υγείας, όπου εντάσσεται αυτός ο τουρισμός σε εθνικές πολιτικές υγείας, θεωρείται κινητήριο δύναμη για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού μέσω της παροχής πρόληψης, ουσιαστικά κάτι κλασικό για τα κέντρα ευεξία, ε, οι αματικέ πηγέ και τον ιατρικό τουρισμό, αντί για θεραπείε εκ των υστέρων. Ε, αν δούμε και τα κέντρα αριστεία, ε, τα δίκτυα αναφορά που έχουν ξεκινήσει τέτοιε ας πούμε για παράδειγμα θεραπείες όλα αυτά τα ειδικευμένα κέντρα τα οποία εργάζονται με συγκεκριμένε ασθένειε, και αυτά θα μπορούσαμε να τα ευθυγραμμίσουμε με τις έννοιες της ε, φιλοξενίας, της μεταφοράς ε, των ξενοδοχειακών υπηρεσιών που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα και τους φίλους για τους συγγενείς των ασθενών. Τέλος, για να κλείσουμε, πρέπει να πούμε ο τουρισμός για λόγους υγείας αντιστοιχεί σε μικρό μερίδιο του συνολικού τουρισμού στην Ευρώπη, 4,3%. Είναι περισσότερο εγχώριος παρά διεθνής και επίσης υπάρχει και μη ιστορικά παρουσία ΣΠΑ κέντρων ιαματικών σε, όλες, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής η ανάπτυξή του και η ποιότητα του βρίσκονται υποπίεση παρότι είναι ήδη υπαρκτέ. Υπάρχουν κάποια ζητήματα με την υλοποίηση τη οδηγία 2011-2024 και τα κόστη θα μπορούσαν να, αντισταθμιστούν με την καλύτερη ολοκλήρωση του τουρισμού ε, για λόγους υγείας και, ε, ε, και των παροχών υγείας. Ως συστάσεις ε, προτείνουμε περισσότερες χρόνες να συμπεριλάβουν ε, της ε, θεραπείας σε ιαματικά κέντρα στις εθνικές τους πολιτικές. Επίσης, στο πλαίσιο της οδηγίας κινητικότητας ε, να αφαιρεθούν οι προκαταβολές διότι οδηγούν σε μη ισορροπημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και επίσης η διάδοση του τουρισμού για την υγεία να λαμβάνεται υπόψη τα στατιστικά στοιχεία και στους TSA και επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο πρόθεση του τουρισμού και το σενάριο ζωτικότητα του τουρισμού για την υγεία να συσταθεί ως ε, αφετηρία για τις ευρωπαϊκές πολιτικές επειδή ενισχύει την υγεία του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτή τη μελέτη. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση και τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους ε, και πρώτα κύριο Σελίβη. Köszönöm szépen, elnök Κύριος Βουέλη, συγγνώμη, έχει το λόγο. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να ζητήσουμε μία έρευνα για το θέμα της, ε, του τουρισμού για λόγους υγείας ε, και να μας παρουσιαστεί αυτό στην ε, Επιτροπή Μεταφορών διότι λίγοι καταλαβαίνουν τι μπορεί να σημάνει αυτό για το μέλλον. στα πλαίσια ε, του κλάδου τουρισμού. Δεν μην επαναλάβω τους αριθμούς. 20 εκατομμύρια εργαζόμενοι ε, που εξαρτώνται από τον τομέα αυτών. Τώρα υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να πούμε οπωσδήποτε εδώ στην Επιτροπή. Οποιαδήποτε έρευνα που αφορά το μέλλον ε, αναφέρει ότι υπάρχουν δύο τομείς όπου σίγουρα θα έχουμε εκρηκτική ανάπτυξη ε, στην επόμενη δεκαετία και στις δύο επόμενες δεκαετίες. Και το βλέπουμε αυτό ήδη. Ο τομέας λοιπόν του τουρισμού και ο τομέας της υγείας. Διότι ε, αυξάνεται η επιθυμία ευημερίας των πολιτών και ευζήν και αφιερώνουν όλο και πιο πολλά ε, χρήματα σε δαπάνες υγείας, ε, υγείας αναζητούν οι άνθρωποι περισσότερες δυνατότητες ε, να νιώσουν καλύτερα και τέτοιου είδους υπηρεσίες σίγουρα θα ζητηθούν και στο μέλλον. Δεν πρέπει δηλαδή να θεωρήσουμε ότι αυτή η έρευνα είναι ένα διοικητικό έγγραφο απλώς. Νομίζω ότι πρέπει να πιάσουμε το σφιγμό της ε, κατάστασης αυτής ε, για να δούμε τι σημαίνει για τους συμπολίτε μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπάρξει λοιπόν ραγδαία ε, άνοδος στον τομέα της υγείας και τον τουρισμό επίσης βέβαια τα ξέρουμε. Ακόμα και αν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μιλάμε για τουρισμό για λόγους υγείας ε, αλλά και από τρίτες χώρες έτσι δηλαδή αν δείτε τον τουρισμό από τη Ρωσία ή ε, τους τουρίστες που έρχονται από την Αραβική Χερσόνησο, ε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλοί που έρχονται εδώ για λόγους υγείας. Και βεβαίως είναι και οι Κινέζοι που ενδιαφέρονται. θα έχουμε μια εκδήλωση για τον τουρισμό και την, ε, τη συνεργασία τουριστικά ζητήματα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας ε, αύριο νομίζω και θα συζητήσει σίγουρα και αυτό το θέμα. Ήθελα λοιπόν να θέσω τα εξής θέματα, τα εξής ε, ερωτήματα. Χρειαζόμαστε μια έκθεση σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου που θα υπογραμμίζει τη σημασία του τουρισμού για λόγους υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που έχει σημασία και για την οικονομία αλλά και για την ευημερία της Ένωσης. Απευθύνομαι λοιπόν στην Πρόεδρο λέγοντας ότι θα ήθελα να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία από την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λυρή. Κύριε Σάντερ, για Σάντερ, τον λόγο. Presidenta, sí, agradecer, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η μελέτη μας δίνει έτσι τροφή προσκέψη για ένα ζήτημα αφενός περίπλοκο και αφετέρου με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σε ό,τι αφορά την οδηγία, εγώ θυμάμαι ότι η οδηγία 2024 δεν είχε ως σκοπό να ενθαρρύνει τον ιατρικό τουρισμό ε, Αντιθέτως, ε, τότε λέγαμε ότι φτιάχνουμε ένα νομικό πλαίσιο που θα διευκολύνει ε, το να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, να βρουν τα φάρμακα ή την περίθαλψη που χρειάζονται εφόσον δεν υπάρχει στη χώρα τους. Και θέλαμε να αντιμετωπίσουμε τον ιατρικό τουρισμό. Διότι ο τουρισμός είναι κάτι που γίνεται έτσι εθελούσια, ενώ η περίθαλψη είναι κάτι το αναγκαίο, είναι μια, μια αναγκαιότητα. Εάν προχωρήσει λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση πρωτοβουλία, κάτι που ε, κάτι με το οποίο συμφωνώ, θα πρέπει να καταστηθεί σαφέ ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο το δικαίωμα, τα δικαιώ, το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να έχουν ε, πρόσβαση σε, σε, ένα καλό ε, σύστημα υγεία στη χώρα του και να μπορούν και να χρησιμοποιήσουν ε, σε πλαισιωμένο τρόπο βεβαίως τα συστήματα υγείας και άλλων κρατομελών ε, όταν δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες τους στη χώρα τους αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι προτεραιότητα για μας ε, να βάλουμε τέλος όπως λέει και η μελέτη στο, στις ε, λίστες αναμονής ε, στην τεφαρή περίθαλψη τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας αυτό πρέπει να είναι σαφές ότι πρόκειται για έναν πολιτικό, ένα πολιτικό ευρωπαϊκό ζήτημα. Τώρα μετά υπάρχει το τουριστικό σκέλος που εντός της προσφοράς της τουριστικής που υπάρχει λαμβάνοντα υπόψη και το ιδιωτικό ενδιαφέρον που υπάρχει, τα ιδιωτικά συμφέροντα αν θέλετε είναι λοιπόν αυτό άλλη μία συνιστόσα ε, της ευημερίας που προσφέρουμε και υπηρεσιών και αυτό πρέπει να ρυθμίζεται και αυτό πρέπει να ελέγχεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα ε, και τις ε, ε, και το κατά αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται και είναι αντικείμενο υπόσχεσης είναι αυτό που λένε ή όχι. τώρα, όταν μιλάμε για μια εθελοντική επιλογή Βεβαίως ε, αυτό μπορεί και να βελτιώνει και την υγεία των προσώπων. Εγώ από την Ισπανία στην δεκαετία του 80, ε, το 70 και του 80, ε, καθώς πλησιάσαμε προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρξε ένα πρόγραμμα στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Υπηρεσιών που μέσω μιας μικρής στήριξης έδινε τη δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν μπορέσει να βγουν από, ε, το, από την πόλη τους, από το χωριό τους ε, που δεν είχαν ποτέ φύγει διακοπές τους δόθηκε η δυνατότητα να μπορούν να πάνε ας πούμε στο Μπενιντόρμ έτσι ε, όχι σε κάποιο εξωτικό μέρος να πάνε στη θάλασσα που δεν είχαν πάει ποτέ ε, με αυτή τη μικρή λοιπόν ενίσχυση δημιουργήθηκε ένα σύστημα το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα και ε, αυτό πραγματικά δημιούργησε πολύ σημαντική ευημερία και μειώθηκε τελικά το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης. Ε, το γεγονός ότι μπορεί να μπορεί κάποιος να ταξιδέψει, ε, να γνωρίσει άλλα, άλλους κόσμους, ε, ε άλλους ανθρώπους, είχαμε και χορούς που οργανώνονταν τότε, είναι μυθική ε, αυτοί οι ηλικιωμένοι άνθρωποι έζησαν τα πάντα ξαφνικά εκεί. Ε, θέλησαμε να το γενικεύσουμε, δεν καταφέραμε να το γενικεύσουμε περαιτέρω, αλλά εν πάση θέλαμε το ίδιο το ταξίδι για ανθρώπους ηλικιωμένους, οικογένειες, να είναι ένας παράγοντας ε, υγείας, ε, ε, ευζοίας και βεβαίως εάν στα πλαίσια αυτής της, ε, του ταξιδιού μπορεί να υπάρχει μια προσφορά να κάνει κάποιος ε, ε να πάει σε κάποια θέρμα ή κάτι τέτοιο στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες ε, οι δραστηριότητες αθλητικές Αυτή η έκθεση πρωτοβουλία λοιπόν θα πρέπει να κάνει αυτό το διαχωρισμό. Ένα πράγμα είναι τα συστήματα υγεία που είναι δικαίωμα πρέπει να, και πρέπει να είναι προσβάσιμα και ποιοτικά και άλλο πράγμα είναι ο τουρισμός. Ως ένας παράγοντας ε, υγείας, ε, ζωίας και μείωση των εξόδων της κοινωνικής ασφάλισης όπως έχει ε, αποδειχθεί σε κάποιες χώρες όπως η δικιά μου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιάλα Σέντερ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μοντέρο. Έχετε το λόγο. Eh, e Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλες και όλους. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν πρόλαβα να ακούσω την παρουσίαση της μελέτης. Ωστόσο, είχα διαβάσει ε, το PowerPoint ε, που μας δόθηκε για τη μελέτη. Από ε, αυτού λοιπόν ήθελα να πω δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι με ικανοποιεί ιδιαίτερα που βρισκόμαστε εδώ στην Επιτροπή μας και κάνουμε αυτή τη συζήτηση που συνδέει τον τουρισμό, την οικονομία και αυτό την οικονομική δραστηριότητα αυτό το τομέα που μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε κάποιες προτεραιότητες δικές μας για τις οικονομίες των κρατών μελών και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο τουριστικός τομέας λοιπόν, ε, οικονομικός τομέας, ε, μπορεί φυσικά να δώσει τη δυνατότητα μέσω της ε, ανταγωνιστικότητας να εξελιχθούν οι τεχνολογίες και να δημιουργήσει εν τέλει έναν σύνδεσμο μεταξύ της διεθνούς διάστασης του τομέα αυτού και του εγχώριου. Έχουν γίνει μελέτες Μια σκέψη για να τροφοδοτήσουμε τη συζήτηση. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε τέτοιου είδους τουρισμός να ενθαρρύνει τις προσπάθειες που γίνεται στον τουριστικό τομέα και στα κράτη ε, μέσω του τουρισμού. Δηλαδή πώς μπορεί αυτός ο τουρισμός να συμπληρώσει άλλους ε, τουριστικούς τομείς. ώστε να καταπολεμηθεί η εποχικότητα του τουρισμού που αποτελεί πρόβλημα να προσελκύει δηλαδή τουρίστες από άλλες χώρες Υπάρχουν φυσικά πολλά και πολύ διαφορετικά συστήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα μπορέσουμε να τα προωθήσουμε, διότι ο καθένας φυσικά θα θέλει να προωθήσει το δικό του σύστημα υγείας. Τίθε βέβαια και ένα θέμα ελέγχων. Ε, πρέπει να γίνει κάποια ανάλυση των διαφόρων συστημάτων υγείας των κρατών μελών ώστε να γίνεται μια θετική, για να το πω έτσι, ε, προώθηση, διαφήμιση τους. Ήθελα να πω και κάτι άλλο ε, για το οποίο είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη. Είναι κάτι που αναφέρεται στη μελέτη. Ε, αναφέρεται η αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας από όπου προέρχομαι και εγώ. Ανήκει στην Πορτογαλία αυτή η περιφέρεια και εκεί υπάρχει ένα κέντρο αριστείας ε, θαλασσοθεραπείας. Γίνεται εκεί δηλαδή τουρισμός για λόγους και ήθελα απλά να επισημάνω αυτό το σημείο το οποίο υπάρχει στη μελέτη. Και Ήθελα να ρωτήσω πώς σε μια άκρος περιφερειακή περιοχή, ε, απομακρυσμένη από γεωγραφική άποψη, παρατηρούμε πώς τέτοιες περιφέρειες ε, μπορούν να υποφεληθούν από κάτι τέτοιο και μπορούν να αποτελέσουν ε, συμπληρωματική αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διάφορες χώρες για να καταπολεμηθεί αυτός ο εποχικός χαρακτήρας, ε, για να δώσουν την ευκαιρία να γίνει περαιτέρω έρευνα στους τομείς της πολιτικής υγείας και του τουρισμού ευεξίας. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι ναι, προφανώς έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση. Το να προετοιμαστούμε για τον τομέα αυτό του τουρισμού που θα συνεχίσει να μεγεθύνεται. Πώς θα προετοιμαστεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει περαιτέρω τον τουρισμό για λόγους υγείας, για λόγους ευεξίας. Ε, ποιοι πόροι είναι αναγκαίοι και πώς θα καταναμηθούν ώστε το τμήμα αυτό της οικονομίας ε, να αξιοποιηθεί επαρκώς και να διδραματίσει τον ρόλο που του αξίζει στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μενίλα, αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Θέλετε να απαντήσετε. Έχετε το λόγο. Okay, on the, on the, first uh, Για το πρώτο ερώτημα. Α, συγγνώμη, δεν σας είδα. Παρακαλώ. Ναι, εντάξει, δεν θα σας το κρατήσω, Πρόεδρε. Καταρχάς να ξεκινήσω επενώντας τον κύριο καθηγητή γιατί τελευταίος έρχεται συχνά, κάνει πολύ καλές παρουσιάσεις για 4,5 λεπτά μάλιστα. Είναι ασυνήθιστο και μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ένας άνθρωπος να μπορεί να περάσει το μήνυμά του. Για το θέμα που συζητούμε τώρα. Το ερώτημα είναι πόσο φιλόδοξοι μπορούμε να είμαστε και πόσο θάρρος πρέπει να δείξουμε για να υπάρξει όντως διαφορά σε έναν ε, τομέα που είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών γιατί Μιλούμε μάλλον για τις δύο πλευρές του ίδιου Ένα είναι η υγεία και τα συστήματα υγείας και το άλλο είναι ο τουρισμός. Οπότε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις φιλοδοξίες μας. Υπάρχει χώρος που μπορεί να καλυφθεί, υπάρχει προσθέμενη αξία που μπορούμε να προσφέρουμε, αλλά αν έχουμε πολύ μεγάλε φιλοδοξίε μπορεί να είμαστε αντιπαραγωγικοί. Να το δούμε τώρα από δύο οπτικές. Καταρχά την υγεία και βεβαίω. ο αρχικός στόχος της παροχής υγείας είναι να φροντίζει την υγεία μας, να αποτρέπει, να θεραπεύει ασθένειες και βεβαίως δεν το αμφισβητώ αυτό καθόλου. Ταυτόχρονα όμως η υγεία είναι ένας τομέας της οικονομίας και ένα κομμάτι του προβλήματος είναι ότι την υγεία δεν την βλέπουμε ως τομέα της οικονομίας. Το κόστος είναι πολύ υψηλό, χωρίς να υπάρχει λόγος πολλές φορές και το αποτέλεσμα καμιά φορά είναι αφισβητήσιμο. Οπότε, αν στο μέλλον και την, ευρω... και την υγεία μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε ως τομέα της υγείας, ως τομέα της οικονομίας, συγγνώμη, τότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, η άλλη οπτική, ο τουρισμός για λόγους υγείας. Δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει, υπάρχει περίπτωση να έχουμε και χώρος να έχουμε αποτελέσματα απέναντι σε τρίτες χώρες. Μιλέστε για την Αραβική Χερσόνησο, τη Ρωσία κλπ. Μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι καλύτερο προς αυτό. Κύριε καθηγητά, μιλήσατε για την ευαισθητοποίηση ε, στις διαφάνειές σας. Νομίζω βέβαια μας δώσατε μάλλον αρκετά αισιόδοξη, αρκετά αισιόδοξα στοιχεία. Αλλά όταν ταξιδεύει κανείς, το ερώτημα είναι πόση προώθηση προϊόντος έχει υποστεί και κατά πόσο μπορεί να, να δει τη διαφορά από κράτος σε κράτος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τρίτα μέρη, τρίτες χώρες προς τα ευρωπαϊκά ΣΠΑ, για παράδειγμα, στα ευρωπαϊκά ιατρικά κέντρα. Γιατί νομίζω ότι κατά κύριο λόγο εθνικός ε, πώ βλέπουμε τα θέματα αυτά. Και επίσης μπορούμε να επενδύσουμε καλύτερα τα κονδύλια μας ως προς αυτό μπορούμε να ταξιδέψουμε σε όλη την Ευρώπη και να βρούμε πάρα πολύ καλά κέντρα ευεξίας, αθλητικά κέντρα, που πολλές φορές χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, αν πάμε σε κάποια από τα σπα αυτά, που μπορεί να είναι και διαμάντια πραγματικά, συχνά ε, αποθαρρύνεται κανείς από το να τα, να, τα, να ταξιδέψει και να πάει σε αυτά γιατί βρίσκονται σε κάποιε ορεινέ περιοχές ε, ή απομακρυσμένες που δεν έχουν τίποτα άλλο να προσφέρουν πέραν του ίδιου του κέντρου. Οπότε έχουμε κάποιο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την επένδυση που κάνουμε σε σύγκριση με τα πρώτης κατηγορίας ε, κέντρα ευεξίας. μήπω μπορούμε να βελτιώσουμε και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ΣΠΑ αυτά. Νομίζω ότι απέναντι στους τρίτου μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και σίγουρα τα κράτη-μέλη μπορούν να επωφεληθούν. Τελευταίο μου σχόλιο για τον τουρισμό πάλι για την υγεία. Εγώ μάλλον είμαι απεσιόδοξος για το κατά πόσο μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προσφέρουμε προσθέμενη αξία. Βεβαίω υπάρχουν ευαισθησίε στο θέμα αυτό, ανά κράτο μέλο, αλλά. Ενθαρρύνουμε τον τουρισμό μεν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι η εθνική θεώρηση των πραγμάτων υπερισχύει. Θα μπορούσαν τα πράγματα ίσως να είναι διαφορετικά με κέντρα αποκατάστασης, ας πούμε. Και επανέρχομαι στο σημείο που έλεγα πριν, ότι η υγεία είναι τομέα τη οικονομία με πολύ ψηλό κόστο. Και πολλέ φορέ χρησιμοποιούμε την ε, θεραπεία γιατί σε εθνικό επίπεδο δεν έχουμε τι δυνατότητες να... ή το κέντρο ευεξία, α πούμε, το σπάτο αντίστοιχο. Οπότε ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε αν θα μπορούσαμε μερικώς να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις θεραπείες από το εθνικό, ε, ε, από το εθνικό προπολογισμό χρησιμοποιώντας όμως τις δυνατότητες των κέντρων ευεξίας ενός άλλου κράτους μέλους. αν έστω σε κάποιο βαθμό δεν μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα της, ε, των ασφαλιών, δεν νομίζω θα τα καταφέρουμε και δεν ξέρω κατά πόσο το είχατε στην ε, παρουσία σας αυτό, νομίζω δεν το είχατε. Αν μπορείτε να το σκεφτείτε θα ήταν καλό μάλλον. Να δώσουμε λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο Σιγητή. Ευχαριστώ. Για το πρώτο σχόλιο, η πρόκληση είναι ότι η μελέτη όντως δεν περιλαμβάνει στοιχεία για Κινέζους, Ρώσους και Άραβες ασθενείς. Οπότε δεν μπορώ να σας δώσω έγκυρα στοιχεία ως προς αυτό. Βεβαίως η ευεξία, η ευημερία είναι πολύ σημαντική ως πτυχή του τουρισμού γιατί δεν μιλούμε μόνο για την υγεία, για τον ιατρικό τουρισμό, αλλά και την ευεξία. Και αυτός, αυτό το είδος τουρισμού αποτελεί έναν πυλώνα. Έτσι απαντώ στο πρώτο ερώτημα. Και συμφωνώ και με αυτό που είπε ο δεύτερος Ευρωβουλευτή. έχουμε από τη μία τα ιατρικά και τα συστήματα υγείας και από την άλλη έχουμε τον τουρισμό, τον τομέα του τουρισμού, το τουριστικό προϊόν και βεβαίω το καλό θα ήταν να υπάρξει κάποιο είδος συνδυασμό. και να πούμε ότι εσείς έχετε ένα ε, ιατρικό κέντρο και σε συνεργασία με ένα ξενοδοχείο ε, θα μπορούσε ο άνθρωπος να μπορεί να παρακολουθεί τη θεραπεία του σε ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον ας πούμε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε πού βρίσκονται αυτές οι καλές πρακτικές και πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα κέντρα αυτά. Πάντα θέλουμε να συνδυάζουμε τους ε, εμπλεκόμενους φορείς και από τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, για το τρίτο ερώτημα, Για τους ανταγωνιστές στον τομέα του τουρισμού και για το ότι ο τουρισμός, η υγεία είναι κλάδος οικονομίας. Ξέρουμε ότι η υγεία και ο τουρισμός είναι όντως ε, θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Αλλά θα μπορούσε να είναι πιθανό ή δυνατό να δούμε και το θέμα των κοινωνικών συστημάτων. Χρειάζεται δηλαδή μια οργάνωση σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο, ανάλογος που βρίσκεται η αρμοδιότητα, για να καθοδηγηθούν σωστά αυτά τα τα τουριστικά προϊόντα σε συνδυασμό με την παροχή ε, υπηρεσιών υγείας έτσι ώστε οι διάφορες περιφέρειες, περιοχές να επικεντρώνονται στην ευημερία, στην ευεξία, στην θεραπεία και των δικών τους βεβαίως πολιτών, αλλά και διεθνών τουριστών που έρχονται. Ίσως αυτό να είναι όντως πρόκληση για να δημιουργήσουμε αυτές τις περιφέρειες υγείας ας πούμε. Και βεβαίως αυτό μάλλον και είναι ένα θέμα της Ευρωπαϊκής ε, να δει πού βρίσκονται οι ευαισθησίες σε θέματα αρμοδιότητας μεταξύ αυτών των περιφερειών, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνδυάσουν τις υπηρεσίες που βρισκονται οι ευαισθησιε σε θεματα αρμοδιοτητας μεταξυ αυτων των περιφερειων ετσι ωστε να μπορεσουν να συνδυασουν τις υπηρεσιες που προσφερουν Και επίσης, για συγκεκριμένες ομάδες στόχους, ηλικιωμένοι για παράδειγμα. Έχουμε ας πούμε τους Βρετανούς πολίτες ως παράδειγμα που πάνε στην Ισπανία για να ζήσουν μόνιμα και χρησιμοποιούν και τις, ε, τα ιατρικά, το σύστημα υγείας της Ισπανίας. Αυτό είναι διαφορετικό βέβαια από το να πάει κανείς να κάνει τις διακοπές του σε ένα κέντρο ευεξίας ε, μέχρι το να πάρει σύνταξη και να μετικήσει σε άλλη χώρα. Ευχαριστούμε για όλες αυτές τις απαντήσεις. Στρέφουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε κάποιο σχόλιο? Κυρία Κρίστινα Μπουρός, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτήν την σημαντική και πολύτιμη μελέτη. Οι πληροφορίες για τη συνεισφορά ε, κάποιων υποτομέων του τουρισμού όπως ο τομέας ε, της υγείας και της ευεξίας ε, δεν είναι πολλές οπότε αυτή η μελέτη έρχεται την κατάλληλη στιγμή σας ευχαριστούμε επίσης για τις συστάσεις όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια σημαντική προσπάθεια για να υποστηρίξει ε, τη διαφοροποίηση των τουριστικών προϊόντων χρησιμοποιώντας ε, και χρήματα από το πρόγραμμα COSME. Εμείς υποστηρίζουμε project τα οποία ε, διευρύνουν την τουριστική σεζόν και παρέχουν και πιο μακροπρόθεσμες θέσεις εργασίας καθώς βεβαίως και την καταπολέμηση της, του υπερβολικού τουρισμού και ο τουρισμός για λόγους υγείας ε, και ευεξίας ε, είναι ε, ένας τρόπος για να συμβεί αυτό. Θα έχουμε το απόγευμα μια μελλοντική παρουσία, πλήρη παρουσίαση για τους στόχους μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο είναι σημαντικό σε σχέση με την παρουσίαση αυτή. Φέτος τα βραβεία που δίδονται για τις ε, καλύτερους προορισμούς θα επικεντρωθούν, θα επικεντρωθούν στα συστήματα τουρισμού για λόγους υγείας. Περιμένουμε συμμετοχή 20 ετών σε αυτό το διαγωνισμό. Ε, θα δώσουμε λοιπόν ένα βραβείο και με αυτό το βραβείο θα αναγνωρίσουμε κάποιους προορισμούς αριστείας ε, που χρησιμοποιούν και που κεφαλοποιούν τον τουρισμό για λόγους υγείας σε διάφορες διάφορους προορισμούς λιγότερο γνωστούς. Αυτή την έκθεση θα την εξετάσουμε λεπτομερώς και θα χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα και τις συστάσεις της δική μας χάραξη πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Μπρούζ για το σύνολο των, της παρέμβασής σας. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ τον κύριο Μενίλκη και τη μελέτη του. Ευχαριστώ που ήρθατε ε, στην Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσετε αυτό το ζήτημα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, συνδέουν το θέμα του τουρισμού, το θέμα της υγείας, αλλά ε, δεν το βλέπει κανείς συχνά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Νομίζω πως είναι σημαντικό για τον ε, τουρισμό για λόγους υγείας ε, να γίνει αυτό κατανοητό να προβληθεί από τους πρόσθελους πολίτες. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος και θα συνεχίσουμε τώρα τις εργασίες μας ε, με την έκθεση της κυρίας Ταπαρντέλ. Κοινοί κανόνες ε, για την εκμετάλλευση των ε, υπηρεσιών αερομεταφορών στην Ένωση. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια και μετά στους κοιόδους εισηγητές. Και βεβαίω και στη συνέχεια θα πάρει λόγο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει το λόγο η συγκεντρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ θετική ενέργεια πριν την ε, ε, παρουσίαση παρουσίασή μου. Εντάξει, με ακούτε. Πολύ ωραία. Ξεκινάω από την αρχή. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, οι ευρωπαϊκές αεραμοταφορές έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Σημαντική ανάπτυξη. Και αυτό βεβαίως συνδέεται και με τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς. Και με βάση αυτήν την ανάπτυξη η ενοικίαση αεροπλάνων με το πλήρωμά τους ε, είναι ένας τρόπος ε, περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου αυτού. Είναι μια πρακτική όλο και πιο διαδεδομένη και αυτό βεβαίως δίνει και μια ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας μιας αεροπορικής εταιρεία. Ορισμένε φορές προκύπτουν τεχνικά προβλήματα, ε, ελλείψεις προσωπικού, αλλά υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να εξεταστούν. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ υπέγραψαν μια διεθνή συμφωνία που προβλέπει απελευθέρωση της αγοράς, της αγοράς δηλαδή της ενοικίασης με πλήρωμα, με πανδρομένων δηλαδή αεροσκαφών. Ε, έκτοτε όμως έχει προταθεί ένας περιορισμός αυτής της φόρμουλας με τρίτες χώρε ε, στα πλαίσια του κανονισμού του 2008. Και εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν το 2017 πρότεινε μια τροποποίηση του άρθρου 13 παράγραφος 3β αυτού του κανονισμού όπου προβλέπεται ε, να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτούς τους περιορισμούς στην ενοικίαση ε, πανδρομένων αεροσκαφών ε, προς τρίτες χώρες όταν ε, αυτή η ενοικίαση εμπίπτει σε μια διεθνή συμφωνία. Είναι μια σύντομη τροποποίηση που παρουσιάζεται ως τεχνική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως ο στόχος είναι να υπάρχει μια συνέπεια σε νομικό επίπεδο μεταξύ του συστήματος αυτού και των ε, ισχύων των διεθνών συμφωνιών. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Όμως ως εισηγήτρια και μετά από συζητήσεις που είχα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τις, ε, τους επαγγελματίες, τις αερομεταφορές, τους εκπροσώπους ε, των ενώσεων για τα δικαιώματα των ταξιδιωτών, νομίζω ότι θα πρέπει να προβούμε σε μια τροποποίηση μια τροποποίηση που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις για τον κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά κριτήρια προστασία των, εργαζομένων αλλά και των ε, ταξιδιωτών. Ανοίγουμε εδώ την ευρωπαϊκή αγορά για την ενοικίαση ε, αεροπλάνων, αεροσκαφών με πλήρωμα κατόπιν διαπραγμάτευσης με την τρίτη χώρα, με την ελόγω τρίτη χώρα. Ε, μπορεί δηλαδή μια δραστηριότητα η οποία είναι προσωρινή να γίνει μόνιμη ε, για να εξασφαλίσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πολίτες, ε, στους ταξιδιώτες. Ε, κατ' εμέ αυτή η ενοικίωση, η ενοικίαση πρέπει να είναι προσωρινή, πρέπει να είναι εξαιρετική. Ε, θα πρέπει να βρούμε ένα σημείο ισορροπίας λοιπόν ανάμεσα στην ανάγκη ευελιξίας για τις εταιρείες αερομεταφορών για να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση και τον σεβασμό των βασικών αρχών που είναι στη βάση λειτουργίας του κλάδου αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι τροπολογίες που έχω προτείνει. Μιλάμε εδώ λοιπόν για ενοικίαση ε, αεροσκαφών για 7 μήνες που μπορεί να παραταθεί για άλλους 7 μήνες εφόσον αποδειχθεί η αναγκαιότητα για κάτι τέτοιο και συνολικά η μέγιστη διάρκεια είναι 14 μήνες. Μπορεί να υπάρξει εξαίρεση εφόσον τα κράτη-μέλη και οι αρχές διαπιστώσουν ε, ότι αιτιολογείται κάτι τέτοιο για να μπορεί να γίνει βεβαίω σεβαστή η βασική αρχή της Ένωσης. Έχουμε λοιπόν προσθέσει εδώ τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, χρειάζεται μια συμφωνία αερομεταφορών ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε λόγο τρίτης χώρας. Δεύτερον, η συμφωνία για την ενοικίαση αεροσκάφου με πλήρωμα ε, θα πρέπει να είναι αμοιβαία και η παράταση της άδειας ενοικίασης θα πρέπει να χορηγείται μόνο αφού μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι για αυτή την περίοδο 14 μηνών η ενοικίαση αεροσκαφών με πλήρωμα έλαβε χώρα ε, με αμοιβαιότητα σε ό,τι αφορά την ε, ισότητα, την ισοτιμία πρόσβαση στην αγορά και βεβαίως οι κανόνες ασφαλείας αλλά και η κοινωνική, τα κοινωνικά κριτήρια αλλά και τα δικαιώματα των εξαιρετών γίνονται σεβαστά. Και η αρμόδια αρχή θα πρέπει επίσης να επαληθεύσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η εν λόγω τρίτη χώρα ε, διέπονται από συγκρίσιμα ε, οικονομικά στοιχεία και υπάρχει ήδη συνεργασία ε, διότι εδώ μιλάμε για την ασφάλεια ε, των αερομεταφορών, την κοινωνική ασφάλεια, τον, την προστασία των ταξιδιωτών και των καρναλωτών. Όταν υπάρχει λοιπόν τέτοια συμφωνία ενοικίωσης, ενοικίωσης αεροσκαφών με τρίτη χώρα, θα πρέπει να φροντίζουμε να υπάρχουν παρεμφερή πρότυπα τα οποία θα ισχύουν για όλους ε, για να μην έχουμε στρεβλώσει στην αγορά για να μην οδηγηθούμε σε κοινωνικό ντάμπινγκ σε αθέμητο ανταγωνισμό θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τον Ιούλιο η Κομισιόν εξέδωσε μια ανακοίνωση όπου προτείνει δύο ακόμα, δύο, δύο ακόμα τροποποιήσεις ό,τι αφορά το δικαίωμα ιδιοκτησίας των, αερο, των εταιριών αερομεταφορών και ε, τα κριτήρια που πρέπει να διέπουν το τη δημόσια υπηρεσία. Μιλάμε λοιπόν εδώ για τρία διαφορετικά κείμενα. Ε, δεν υπάρχει ε, επαρκή νομική σαφήνεια όμως. Χρειαζόμαστε λοιπόν πρώτα μια μελέτη αντικτύπου με επιχειρήματα για μια τέτοια τροποποίηση και από εκεί πέρα να δούμε εάν ο κανονισμός θα πρέπει να τροποποιηθεί ή όχι. Από εκεί πέρα αναμένω να ακούσω τις απόψεις ε, των συναδέλφων, των σχεδόν εισηγητών και το τελευταίο που ήθελα να πω και να θυμίσω είναι ότι θα ήθελα εγώ να επιδείξω ανοιχτό πνεύμα είμαι έτοιμη να ακούσω όλα τα επιχειρήματα θέλουμε να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ αφενός του ανοίγματο της αγοράς αλλά αφετέρου και των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απέναντι στους αδέλφους. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ την κυρία Ταπαρντέλ. Θα ξεκινήσει αμέσως η συζήτηση και θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκέλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Ακούσαμε ποιο είναι το σημείο κίνησης. Είπα και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν την συμφωνία του 2007 για τις αεροπορικές εταιρείες που μπορούν να, κάνουν, να συνάπτουν τέτοιες συμβάσεις ε, χωρίς περιορισμούς. Έχουμε κάποιους περιορισμούς ήδη από το 2008 με τη σχετική νομοθεσία και η ΕΠΑ από τότε ζητούν διευκρινήσεις. Και αυτό θα γίνει, λέει η Κομισιόν, μέσω μιας συγκεκριμένης και ρεαλιστικής προσθήκης στο 13.3 του κανονισμού. Βεβαίω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν ασχολούμαστε με τέτοια ευαίσθητα δεδομένα για τις ε, συμφωνίες αυτές και τη Συμφωνία Βάσης Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα. Αυτή είναι η μόνη ε, παρέκκληση που μπορεί να υπάρξει από το 13.3. Ένα σημείο είναι αυτό. Η Συμφωνία για τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες ΕΕ λαμβάνει υπόψη τις περαιτέρω νομοθεσίες που υπάρχουν σχετικά στο Ενατιλογική ε, Σκέψη 8 και όπως αναφέρθηκε στο 13.3 του 2008 του 2008. Ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να δεχτώ τις προτάσεις σας. Τροπολογία 1. Κατά τη δική μας άποψη, για την αρμόδια αρχή αδειοδότησης ε, επιβάλλει καθήκοντα που δεν μπορεί να τα επομιστεί. Γιατί μιλούμε για παρέμβαση στην νομοθεσία τρίτων χωρών. Και επίσης θα πρέπει να είναι, λέει, συγκρίσιμες νομικά αυτές οι διατάξεις με το ευρωπαϊκό δίκαιο και με τα δίκαια των κρατών μελών. Και μετά αυτές οι διαφορές θα πρέπει να σταθμιστούν με κάποια δικαιώματα προστασίας για τα θεωρητικά ε, συμφέροντα κάποιων πιθανών ταξιδιωτών. Ε, μιλούμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο όμως θα κερδίσουμε κάτι μέσω αυτής της ε, νέας συμφωνίας. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ πρακτικό αυτό που προτείνεται. Τροπολογία 2. Επίσης μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένη ώστε να υπάρξει αυτή η επιθυμητή διευκρίνηση για τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Και Απέναντι σε αυτές τις ε, ισχύουσες διατάξεις ισχύει ε, μερικώς το 13.3. Γιατί ούτως ή άλλως είναι θέμα ευθύνης της αεροπορικής εταιρεία και της αβιβαιότητας που επιθυμείται να επιτευχθεί από την Συμφωνία ΕΕ ΕΠΑ. ΕΕ. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχτώ τις προτάσεις σας κυρία Συγήτρια. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φώστερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά ευχαριστώ στην Κλάδια Ταπαρντάλ για τις ε, έντονες προσπάθειές της και για τις πολύ καλές της ε, επεξηγήσεις. Κατά την απόψή μου, η πρόταση της Κομισιόν είναι καλή και επαρκής. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι διότι αν πάμε πίσω στο 1992 στο ΙΚΑΚ 21 καθώς 1 όλοι τότε ε, συμμορφωθήκαμε με τους κανόνες ε, για το dry leasing και το wet dump. Ε, υπήρχαν και διεθνείς συμφωνίες διότι ναι, γινόταν μίσθωση αεροσκαφών από τρίτε χώρε και αντίστροφα νομίζω η Air France ε, είχε μισθώσει σε κάποια εταιρεία στο Νοτιοειρηνικό. Ε, δεν ξέρω πώ ακριβώ το έκαναν βάσει ποιων πραγμάτων, αλλά είμαι σίγουρη ότι ήταν επιτυχέ το εγχείρημα. Δεν είναι λοιπόν κάποια πρακτική νέα. Από δική μου εμπειρία προσωπικά, όταν δούλευα στην British Airways, είχαμε κάποια προβλήματα συντήρηση στο στόλο και χρειάστηκε να μισθώσουμε αεροσκάφη από την Τρανσάβια που είναι Ολλανδική εταιρεία για πάνω από δύο χρόνια. Διότι για να γίνει βάθμιση του στόλου που είχαν, διότι ήταν τεράστιο ο στόλο ήταν αδύνατο αυτό να γίνει σε 7 και σε 14 μήνες, οπότε ήταν ε, πολύ καλή συμφωνία. Ήταν ένα μείγμα αεροσκαφών, πληρωμάτων κτλ. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε καλά πριν να θέσουμε χρονικούς περιορισμούς σε κάτι τέτοιο ε, θέματα. Διότι ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις θα είναι ένα-δυο μήνες. Και ξέρετε δεν είναι κάτι φθηνό. Ε, και υπάρχει ένας μύθος ότι αν οι εταιρείε αποφασίζουν ε, ότι δεν έχουν αρκετό πλήρωμα και αεροσκάφη θα αρχίσουν να μισθώνουν για πάντα. Αυτό είναι μύθος. Είναι ανακριβές. Μισθώνουν αεροσκάφη μόνο όταν το χρειάζονται για συγκεκριμένους λόγους. Οπότε εγώ θα έλεγα να μην το περιορίσουμε χρονικά. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω όσον αφορά τις κοινωνικές συνθήκες και την νομοθεσία για την απασχόληση. Κανείς δεν λέει να έχουμε ανεπαρκείς κοινωνικές συνθήκες. Αλλά το να θεωρούμε δεδομένο ότι οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών απασχολούν ανθρώπους υπό φρικτές συνθήκες είναι αρκετά λαζονικό θεωρώ. Διότι πολύ συχνά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όλοι πρέπει να συμμορφώνονται με την νομοθεσία σε όλους τους τομείς. Ε, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε η Lufthansa έχει μια κινέζικη εταιρεία στην ε, ε, αεροπορική συμμαχία και αν θέλει να μισθώσει από εκεί θα ζητήσει τι αντίγραφο όλης της νομοθεσίας για την απασχόληση στην Κίνα Οπότε πρέπει να είμαστε κάπω λογικοί, να μην είμαστε υπερβολικά περιοριστικοί στα όσα λέμε εδώ, διότι αυτό ο αρωματοφορέας ε, είμαι βέβαιος ότι είναι αξιόλογος και ότι απασχολεί ανθρώπους ε, βάσει όλων των απαιτήσεων που επιθυμεί και η Λουφθάνσα. Συνολικά πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να προσέξουμε, όπως είπε και ο κ. Γκάλαν, να προσέχουμε λοιπόν τι θα βάλουμε μέσα στο κείμενο γιατί δεν θέλουμε να το περιπλέξουμε υπερβολικά για λάθος λόγους. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά την κυρία Ταπαρντέλ. Ευχαριστούμε κυρία Μπελμπάου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω και την κυρία Ταπαρντέλ, τη συνάδελφο για το έργο της. Εγώ νομίζω ότι δεν θα εκπλαγείτε αυτό που θα, γι αυτό που θα πω, με αυτό που θα πω. Θα είμαι και σύντομη. Είναι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τεχνικής υφής. Εμείς οι φιλελεύθεροι δεν θεωρούμε ότι πρέπει τώρα να διευρύνουμε το περιεχόμενο αυτή της πρότασης. Προτιμούμε μια γρήγορη επίλυση αυτού του ζητήματος, του τεχνικού, και αν χρειαστεί η αναθεώρηση να κάνουμε μια αναθεώρηση. Βεβαίω αυτό να γίνει με συνένεση και με σύνεση. Η κυρία Ταπαντέλ γνωρίζει τη θέση μας εδώ και πολύ καιρό και εμείς ως πολιτική ομάδα θεωρούμε ότι ε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε θέση από αυτού. Θα ήταν καλό να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν προβλέπει κάποια αναθεώρηση. Πότε και πότε διότι πολλά από αυτά που είπε η κυρία Ταπαντέλ ε, για μας δεν τίθενται. Ε, φυσικά και είναι σημαντικά. Ε, θέλουμε έναν ισχυρό καινοτόμο κλάδο, να προστατεύουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα δικαιώματα των ταξιδιωτών. Αυτά είναι αισθήματα τα οποία, με τα οποία συμφωνούμε. Το βασικό όμω είναι συμφωνούμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα τεχνικό θέμα και προχωράμε ή θέλουμε να το ανοίξουμε, να το διαβρύνουμε. Εμεί δεν θέλουμε να το διαβρύνουμε. Θέλουμε να επιληθεί αυτό το τεχνικό ζήτημα άμεσα. Um, Ευχαριστώ. Καλωσορίζω την προσεκτική προσέγγιση της συναδέλφου Ταπαρδέλ. Δεν συμφωνώ όμως ότι είναι μόνο τεχνικό θέμα. Είναι πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα που θα έχει πολύ αρνητικές συνέπειες και δεν συμφωνώ με την Τζάκι Φώστερ. Κυρίως, ε, τι έκπληξη βέβαια, Κυρίω αν σκεφτούμε πέρσι τον Ιούλιο το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε έγκριση στις, ε, στις ε, βρετανικές αερογραμμές να μισθώσουν αρκετά ε, αεροσκάφη και πραγματικά έγιναν πάρα πολλέ παρατηρήσει και υπήρξε πάρα πολλή συζήτηση ω προ αυτό. Η Επιτροπή Τραν προσπάθησε να υποβάλει μια προφορική ερώτηση στην Ολομέλη και δυστυχώ άλλε ομάδε μα μπλόκαραν. Οπότε θα ήθελα να το θέσω αυτό. Και για τα θέματα που συζητούμε, Βεβαίω υπάρχουν μεγάλε ανησυχίε για τι διατάξει για την ασφάλεια και την υγεία και τι απαιτήσει από τι ε, ε, αεροπορικέ γραμμέ του Κατάρ, α πούμε, για την μεταχείριση των γυναικών, ε, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα παράδειγμα είναι αυτό ποια είναι ότι η ε, μίσθωση τέτοιων αεροσκάφων, αεροσκαφών μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολύ αρνητικό τρόπο. Δεν λέω ότι πάντα γίνεται αυτό, αλλά γίνεται. Και επίση η αμοιβαιότητα που είπε και η συνάδελφο. Αν δούμε τον κώδικα τη ε, FAA, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι περιορισμοί για την μίσθωση τέτοιων αεροσκαφών. Και θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν αν το έχει μελετήσει ε, σωστά για την αμοιβαιότητα σε τέτοιου είδου συμφωνίε και συμβάσει. Γιατί εδώ έχουμε και μερικώ ε, ε, ε, θέματα που άπτονται και του καμποτάζ και θέματα που άπτονται και τη ασφάλεια. Οπότε θα πρέπει μάλλον να γίνει μια γενική αναθεώρηση. Άρα, γιατί το κάνουμε τώρα αυτό, εφόσον δεν έχει υπάρξει ακόμα αξιολόγηση αντικτύπου. Και επίση η Κομισιόν μπορεί να σχολιάσει την έκθεση τη Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που ήταν πάρα πολύ αρνητική. Ε, δέχτηκαν ότι μάλλον θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση, αλλά είπαν ότι χρειάζονται περισσότερε διευκρινήσει. Και μα ανησυχεί επίσης το θέμα της κατάχρησης των προτύπων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και επίσης πιο γενικά να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτός ο πολύ ωραίος κοινωνικό πυλώνα για τις αεροπορικές μεταφορές που μας τον υπεσχεθήκατε και σε εμά και, στην, και στις επιχειρήσεις, πού είναι για να υπάρξει αυτή η σωστή εταιρική σχέση για του εμπλεκόμενου φορεί στην αεροπορία, γιατί ακόμα δεν την έχουμε δει και δεν θα πρέπει να μας ζητάτε να κάνουμε τεχνικές αλλαγές σε ένα κείμενο τέτοιο όταν δεν υπάρχει σωστή και γενικότερη, συνολικότερη προσέγγιση για την αεροπλοεία. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν είχα βαθύνει επί του αυτού, αλλά βλέποντας εδώ τις προτάσεις ε, τροποποίησης της κυρίας Ταπαρντέλ, εγώ συμφωνώ μαζί της ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλά προτείνει μια τεχνική αλλαγή. Βεβαίω ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για αμυγό τεχνικά ζητήματα πάντα κρύβονται ε, κοινωνικά ζητήματα ε, τα οποία δεν φαίνονται στην επιφάνεια. Εάν λοιπόν δεν προβλέπετε κάποια αναθεώρηση με ένα κοινωνικό πυλώνα, τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στην πρόταση της κυρίας Ταπαρντέλ διότι παράλληλα εξετάζουμε το πακέτο ε, για τις οδικές μεταφορές όπου κάθε φορτίγατζης ε, θα πρέπει να ακολουθεί διάφορες συμβάσεις, διάφορες νόρμες ε, και των επτά χωρών μελών που θα διασχίσει στις αερομεταφορές είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε όμως ενοικίαση με πλήρωμα προς οποιαδήποτε τρίτη χώρα ε, με οποιαδήποτε νομοθεσία κοινωνική, για να μην πούμε την περιβαλλοντική. Ε, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ε, δεν είναι ένα αμυγός τεχνικό ζήτημα, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και να πούμε τουλάχιστον στην Κομισιόν ότι είναι αναγκαίο αυτές οι πτυχές να αντιμετωπιστούν. Ο κοινωνικός αντίκτυπος αλλά και άλλοι αντίκτυποι στον τομέα των αερομεταφορών. Και κάτι άλλο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, αυτή η, η φόρμουλα, η light, όπου κάθε, κάθε εταιρεία θα μπορεί ε, να νοικιάζει αυτοκίνητα όπου θέλει και με το πλήρωμα που θέλει. Ε, ε, όλα γίνονται την, ε, με βάση την διευκόλυνση, την ευελιξία, την ε, ταχύτητα. Δεν πρέπει να οδηγηθούμε όμως και σε ένα Uber στον τομέα των αερομεταφορών. Αν υπάρχει μια πλατφόρμα δηλαδή ε, που θα προσφέρει στον τομέα του τουρισμού διάφορες τέτοιου υπηρεσίε. να ανοίξουμε λέει, τη δυνατότητα μέσω μιας πλατφόρμας ε, να μπορούμε να υπογράφουμε συμβάσεις ενοικίασης ε, αεροσκαφών με πλήρωματα από τρίτες χώρες. Ε. Αυτά είναι κάπως προβληματικά σε ό,τι το πλαίσιο που θέλουμε. Ευχαριστώ την κυρία Γιάλα Σέντερ. Απευθύνομαι τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Κορνέλης, καλή σας μέρα. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την συγγέντρια την κυρία Ταπαρντέλα για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει για το θέμα αυτό και ευχαριστώ επίσης όλους τους υπόλοιπους για την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων σήμερα το πρωί. Πραγματικά αγγίζει το πυρήνα όλων των ζητημάτων που προκύπτουν στον τομέα αυτών. Να θυμηθούμε για ένα λεπτό από πού προέρχεται αυτή η πρόθεση της Κομισιόν. Όπως πολύ, η ε, πρόθεσή της είναι να ευθυγραμμίσει την νομοθεσία μας ε, μετά όσα πρέπει να κάνουμε ως αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης συμφωνίας για την αεροπορία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόθεση δεν ήταν να αλλάξουμε την προσέγγιση της μίσθωσης γενικότερα, ούτε εσωτερικά, ούτε με τις τρίτες χώρες. Ε, δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση να ανοίξουμε την πόρτα σε περαιτέρω απελευθέρωση σε σχέση με άλλες χώρες, τρίτες χώρες. Απλά σκοπός ήταν να ευθυγραμμιστούμε με τις υπάρχουσες ε, διεθνείς συμφωνίες, ε, ειδικότερα με τις ΗΠΑ. Και όπως είπαν μερικοί από εσά, πρόκειται για μια τεχνική, νομοθετική, νομική ουσιαστικά ευθυγράμμιση. Αυτό προτείνουμε εδώ. Αυτό παρατηρούμε είναι το κείμενο του σχεδίου έκθεσης φαίνεται να επιτρέπει ένα ευρύτερο πλαίσιο, πιο ανοιχτό για ε, πλήρη εκμίστοση για wet list με τρίτες χώρες. Παρότι προτείνονται πολλές νέες συνθήκες στην έκθεση. Αυτό υπερβαίνει τις προθέσεις της Επιτροπής στην αρχική της πρόταση, όπου προέβλεπε απλή νομική ευθυγράμμιση ώστε να καλυφθεί η συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ο κινδύνος είναι η έκθεση και οι τροπολογίες που προτείνει η συγγήτρια να μας εμποδίσουν από το να προχωρήσουμε στην εκπλήρωση των σημερινών μας υποχρεώσεων ενώπιον των ΗΠΑ. Τώρα, πιο γενικά, τα ζητήματα που αναφέρθηκαν πράγματι είναι σημαντικά ζητήματα. Εμείς ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με αναθεώρηση του βασικού κανονισμού της εσωτερικής αγοράς 2008 ε, του 2008 που συμπεριλαμβάνει και το ζήτημα του wet leasing και πιστεύουμε ότι αυτό το έργο που έχει ξεκινήσει τώρα με την αξιολόγηση του υπάρχοντος κανονισμού και που θα συνεχιστεί με μια σωστή και πλήρη εκτίμηση αντικτύπου όλα αυτά θα δημιουργήσουν το πλαίσιο φέτος και του χρόνου ώστε να ακολουθήσει μια πλήρη συζήτηση για τις ε, συμφωνίες wet leasing στην εσωτερική μας αγορά και τους όρους από τους οποίους πρέπει να ε, συνάπτονται. Είναι σημα... σαφές ότι το wet leasing είναι μια σημαντική πτυχή της αεροπορικής βιομηχανίας ε, η οποία δεν μπορεί να μην το χρησιμοποιεί δεν είναι μόνο κάτι που κάνουν ξένοι αερομεταφορείς στις δικές μας χώρες και εμείς μισθώνουμε αεροσκάφη σε τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα όμως το wet leasing δεν πρέπει να δημιουργεί στρέβλωση του ανταγωνισμού ούτε να υπονομεύει τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν στην ευρωπαϊκή και στην εσωτερική αγορά. Πιστεύω σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι. Αυτό που θέλουμε να εξετάσουμε στην αναθεώρηση αυτή του κανονισμού 1008 του 2008 θα είναι το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τη σωστή χρήση του List ε, προς όφελος των επιβατών και των αερομεταφορέων χωρίς να δημιουργείται στρέβλωση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς. Τώρα, για να πάμε στις απαρχέ αυτής της πρότασης. Για να συνδεθεί μια συγκεκριμένη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ για το wet leasing, οι διαπραγματεύσει σημείωσαν καλή εξέλιξη και έτσι καταφέραμε να παρουσιάσουμε το σχέδιο συμφωνία στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι δημόσιο το έγγραφο αυτό, δεν έχει δημοσιοποιηθεί διότι οι διαπραγματεύσει δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ωστόσο όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου μπορούν να έχουν πρόσβαση στο κείμενο αυτό για να δουν το περιεχόμενό του. Εκεί λοιπόν μπορείτε να δείτε ότι αυτή η νέα συμφωνία ε, wet leasing με τις ΗΠΑ, Πολιτείες θα περιορίζεται σε δραστηριότητες των Αμερικανών αερομεταφορέων που ήδη ε, πραγματοποιούν εντός της Ευρώπης. Δεν δημιουργούμε δηλαδή ευρύτερη πρόσβαση στην αγορά μας με αυτή τη συμφωνία. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτού του τύπου το wet list δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των επιβατών. Τα δικαιώματα των επιβατών παραμένουν απολύτω τα ίδια. Είτε πετάτε με μια ευρωπαϊκή εταιρεία, είτε με, με ένα αεροπλάνο μισθωμένο από αμερικανική εταιρεία μέσω wet list. Θα παρατηρηστεί λοιπόν ότι το σχέδιο αυτό συμφωνία αναφέρεται στι αρχέ που περιλαμβάνονται στη γενική μα συμφωνία Open Skies με τι ΗΠΑ ε, σε θέματα ανταγωνισμού και σεβασμού των εκατέρωθεν κανόνων και κανονισμών. Ε, σεβασμού δηλαδή των κανόνων της χώρας όπου ε, πετάει κανείς. Ε, και αυτό επηρεάζει φυσικά και τις πτήσεις wet στην Ευρώπη. Χαιρόμαστε λοιπόν μάλιστα που υπάρχει μια ενημέρωση μεταξύ μας και για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις και με τα μέλη του Κοινοβουλίου ώστε να διασφαλίσουμε ότι το κείμενο αυτό δεν θα ανοίξει πόρτες ανεπιθύμητες. Σε γενικέ γραμμέ πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το wet list και το ρόλο του και τι συνθήκε υπό τι οποίε υλοποιείται στο πλαίσιο τη αναθεώρηση του κανονισμού 2008, του 2008. Ε, πρότασή μα είναι, εφόσον ε, προκύψουν ανησυχίε στο Κοινοβούλιο για αυτή την τεχνική, νομική ε, τροποποίηση που φοβάστε ότι μπορεί να ανοίξει κάποια ενδεχόμενα, κάποιε δυνατότητε που δεν συμβαίνει φυσικά αυτό, αλλά σε περίπτωση που υπάρχουν ανησυχίε, αν θέλετε να ενισχύσουμε ή να περιορίσουμε την τροποποίηση, αυτό μπορεί να γίνει ώστε να είναι σαφέ ότι καλύπτει μόνο τη συμφωνία με τι ΗΠΑ. Είτε με άμεση αναφορά στον τίτλο τη συμφωνία, είτε με την εισαγωγή κάποιου σημερομηνία. Ε, ε, λήξη ή κάποια αναφορά συμμόρφωση με τις υπάρχουσες διεθνεί υποχρεώσεις μας όπου φυσικά θα εφαρμόζεται μόνο στι περιπτώσεις όπου έχουμε ήδη μία ε, πλήρη συμφωνία. Αυτό έχω να προτείνω εγώ για το μέλλον, ώστε να καθησυχάσουμε τις ανησυχίες, να περιορίσουμε το κείμενο και όχι να συμπεριλάβουμε μία ευρεία νέα προσέγγιση για το wet lease ε, όσον αφορά τις τρίτες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κορνελής. Κύριε Ταπαρντέλ, για να κλείσουμε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχήν να ευχαριστήσω τους ε, συνεισηγητές ε, για τις απόψεις τους. Ε, συνεργαστήκαμε εδώ στην Επιτροπή Τραν για διάφορα ζητήματα. Γνωρίζουν ότι είμαι ανοιχτή, ότι δείχνω κατανόηση και ότι βεβαίως αυτό που θέλω είναι όπως και αυτή να έχουμε μια καλή νομοθεσία για τους ε, συμπολίτες μας. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Είμαι βέβαιη ότι θα φτάσουμε σε ένα πολύ καλό κείμενο. Είμαι ανοιχτή προς τις τροπολογίες. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα πεδίο ίσου ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά που θα εξασφαλίζει όμως και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των ταξιδιωτών σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι το γνωρίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Η παρουσίαση έγινε εδώ στο Κοινοβούλιο καθυστερημένα, ακριβώς για να έχουμε και το χρόνο να εντοπίσουμε κάποια λύση και να δώσουμε τη δυνατότητα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει τι καλύτερες δυνατές λύσεις για την ε, επίλυση των ζητημάτων αυτών ε, τα οποία η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι αμυγό τεχνικά. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του συναδέλφου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, Βεβαίω μπορεί να είναι αμυγό τεχνικό το ζήτημα με βάση τις διαπραγματεύσει με τους Αμερικανούς όμως οι διαπραγματεύσει ε, σε τεχνικό επίπεδο είναι στι αρμοδιότητε τη Κομισιόν προφανώς αλλά το Κοινοβούλιο είναι υποχρεωμένο να μπορέσει να ψηφίσει μια σωστή νομοθεσία. Ε, είναι δική μας αρμοδιότητα θέμα αυτό. Εξού και η πρότασή μου για μια έκθεση. Βεβαίως ε, αναφερθήκατε στο γεγονός ότι θέλετε να επιλύσετε ένα τεχνικό ζήτημα στις σχέσεις μας με τους Αμερικανούς. Πολύ ωραία. Να σας θυμίσω όμως ότι αυτή η τεχνική πρόταση που έχετε υποβάλει πουθενά δεν λέει ότι μιλάμε απλά για μια διμερή ε, σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πολιτειών. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ως ε, Ευρωβουλευτής ε, πρέπει να εξασφαλίσω ότι εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή αγορά σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες με τρίτες χώρες, με όλες τις τρίτες χώρες. Δεν ε, μιλάμε εδώ για μη σεβασμό συμφωνιών, ούτε θέλουμε να ανοίξουμε παντελώ την αγορά μα. Απευθυνόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι εσεί διαπραγματεύεστε αυτέ τι συμφωνίε και εμεί απλά τι εγκρίνουμε εκ των υστέρων συχνά χωρίς να έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Εσείς όμως, ε, ως διαπραγματευτής της Ένωσης, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την υποχρέωση να πραγματεύεται σωστές συμφωνίες, χωρίς ε, να ε, θυσιάζουμε τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και τις ευρωπαϊκές αρχές. Ε, δεν νομίζω να υπάρχει κανείς εδώ που να θέλει μια συμφωνία με τους Αμερικανούς που δεν θα σέβεται μια σειρά από αρχές, ε, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των ταξιδιωτών, ε, τον θεμητό ανταγωνισμό και βεβαίω την ανάγκη να δώσουμε στις ευρωπαϊκές εταιρείες τη δυνατότητα να απαντήσουν Ε, στα, στο αιτή, στα αιτήματα που υπάρχουν, στις ανάγκες που υπάρχουν στο τομέα του τουρισμού. Ανοίγουμε λοιπόν εδώ ένα διάλογο για να δώσουμε και στους πολίτες αλλά και στις αερομεταφορές, ε, στις εταιρείες αερομεταφορών να δώσουν με τη δυνατότητα να προστατευτούν τα δικαιώματα όλων. Θα ήθελα βεβαίως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει μια μελέτη αντικτύπου Συζητούμε όμως εδώ πάνω από έξι μήνες και εξακολουθούμε να είμαστε στη φάση αξιολόγησης. Θα προτιμούσα να υπήρχε μεγαλύτερη φιλοδοξία, ε, διότι αυτό θα έχει πτώσει για το σύνολο των αερομεταφορών. Ευχαριστώ κυρία Εισηγήτρια, κυρία Ταπαντέλ, να θυμίσω ότι 16 Μαρτίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ναι, κυρία Άντερσον, θέλετε κάτι. Ναι, ήθελα απλώ να πω για την προφορική ερώτηση που έχει μπλοκαριστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων για το leasing. Μπορείτε να το ξαναθέσετε παρακαλώ το θέμα αυτό στη διάσκεψη των Προέδρων, διότι ε, είναι ένα θέμα που μα ανησυχεί ιδιαίτερα ε, και υπάρχουν εκεί μεγάλε δυνατότητε καταχρήσεων. Ναι, θα είναι στη μεσή διάταξη τη συνεδρία των συντονιστών, κύριε Άντερσον. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, επειδή έκανα ένα λάθο προηγουμένω. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 16 Μαρτίου, όχι στις 5 το απόγευμα, αλλά στις 11 το πρωί. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας για σήμερα το πρωί. Θα τα ξαναπούμε στις 5, λέει, πρόεδρος 3 εννοεί, στις 3. Στις 3 ε, την Task Force για τον τουρισμό και το έτος τουρισμού μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ε, ευχαριστώ, θα τα πούμε το απόγευμα.